και να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 Καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα ε, και μέχρι ότου έρθουν και ε, κάποια μέλη από κάποιες πολιτικές ομάδες. Τουλάχιστον νομίζω ότι οι κυριότεροι είμαστε παρόντες, οι κυριότερες ομάδες. Χαίρομαι πολύ σήμερα το πρωί που μπορώ να εισαγάγω σε σας να τον παρουσιάσω και να τον καλωσορίσω τον κύριο Γκάριγκες, τον πρόεδρο το, της υπηρεσίας ε, Future Trade Commission από της ΗΠΑ, φυσικά του αρμόδιου ρυθμιστικού οργάνου της ΗΠΑ για ένα μεγάλο τμήμα των παραγόγων, της αγοράς παραγόγων της ΗΠΑ. Και ο κύριος Γκένσλερ θα μας δώσει μια εισαγωγική, μια εισαγωγή και Νομίζω είχαμε και διανομή, θα διανεμηθούν και τα αντίτυπα της παρέμβασής του. Δεν είναι βέβαιο ότι θα εκφωνήσει λόγο που θα παραμείνει πιστός σε αυτό το κείμενο. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μετά από την παρέμβασή του θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που είσαστε εδώ και μπορείτε να μας παρουσιάσετε κάποια από τα τεκτενόμενα στη ΣΥΠΑ και να μας βοηθήσετε ίσως κιόλας να και εμείς να προσθέσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το σημαντικό τομέα της ρύθμισης του τομέα παραγωγών. Έχετε τον λόγο. Σε καλημέρα σας. There uh, Good morning. Uh, Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας, Πρόεδρε, μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να μιλήσουμε για τα παράγωγα, την αγορά παραγωγών και τα swaps. Θα ήθελα να παρουσιάσω τις δύο μου κόρες, την Λί και την που είναι παρούσες εδώ και που έχουν και τις ε, διακοπές τους, αρινές ε, διακοπές και αποφάσισαν να έρθουν μαζί μου και αυτές ε, εδώ. Η κρίση του 2008, η χρηματοοικονομική αυτή κρίση, ήταν παγκόσμια φυσικά και το χρηματοοικονομικό σύστημα πιστεύω απέτυχε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και το ρυθμιστικό σύστημα του χρηματοπιστωτικού οικονομικού τομέα απέτυχε κάποιοι στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ που ποτέ δεν είχαν κάποια σύνδεση με παράγωγα ή κάποια άλλα τέτοια ωραία συμβόλαια οικονομικά επλήγησαν πάμπολοι άνθρωποι από τις πράξεις όσων εμπλεκόντουσαν σε σχέση με τα παράγωγα που ήταν στο επίκεντρο του 2008 και της κρίσης προσέθεσαν μοχλική δύναμη και δημιουργούσαν μεγαλύτερο κίνητο με μικρότερα κεφάλαια. Φυσικά σώθηκε η AIG με 180 δις δολάρια από την κυβέρνηση των ε, ΗΠΑ όταν είχαμε 2-3 ε, εκατομμύρια παραγόγων που ε, διαχειριζόντουσαν και από πλευράς Λονδίνου. Όμως ε, στο παγκόσμιο σύστημα ήταν συνδεδεμένο όλο αυτό το σύστημα και σχεδόν κατέρευσε το παγκόσμιο σύστημα μετά. Όπως ακούσαμε, πολλά από τα χρήματα μέσω της AIG, χρήματα φορολογουμένων της ΕΠΑ, περνούσαν μέσω των ε, διεθνών τραπεζών παγκόσμια. Όλα αυτά δείχνουν ότι πως ε, αυτές οι άτακτε συναλλαγέ οδήγησαν στο να αυξηθεί ο κίνδυνο για του πολίτε. Τούτου είδους οι συναλλαγές δεν έχουν γεωγραφικά όρια. Η σημερινή αγορά απαιτεί μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση ρυθμιστικά θα χρειαζόμαστε και εργαζόμαστε πολύ στενά όλοι μας ε, για αυτό το στόχο και ευχαριστώ την Πρόεδρο που με προσκάλεσε να δημιουργήσουμε αυτό το συντονιστικό πλαίσιο. Προτού αναφερθώ στις μεταρρυθμίσεις και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τις ρυθμιστικές προσπάθειες της ΕΠΑ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρηματοοικονομικής κρίσης 1930 πήγε ο Πρόεδρος Ρούσβελτ και ζήτησε να υπάρξει κάλυψη των ασφαλιστικών ε, συμβολέων, Exchange Commission, και την άλλη πράξη που ζήτησε νομοθετικά να ρυθμιστεί σε σχέση με το On Exchange Futures και σε σχέση με τα σιτηρά για παράδειγμα, σίτο, κρυθάρι και τα λοιπά και τις, ε, τα γεωργικά αγαθά. Αυτή είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και υπό αυτή την ε, ρυθμιστική ιδιότητα ομιλώ σήμερα. Στην Επιτροπή μας ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ελεύθερες δίκαιες αγορές, ελεύθερες από καταχρήσεις και στρεβλώσεις. Και βλέπουμε ότι τα, ε, οι ρυθμιστές ε, από πλευράς μας όσον αφορά ε, τους συμψηφισμούς και τις συναλλαγές πρέπει να βαίνουν καλώς. Ε, και επίσης επιτηρούμε την αγορά, να διασφαλίσουμε ότι όλοι συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις. Τώρα παράγωγα και καινοτομία, πράγμα που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και από τους ε, ε, προγόνους μας το 1930 αριθμίστηκε και με μεγάλη αλλαγή το 1980. Αυτή η αλλαγή είναι η αλλαγή του over-the-counter derivatives. Αυτά τα παράγωγα όπως τα αποκαλούμε δεν παίρνανε μέσω από χρηματιστήρια και δεν ρυθμιζόντουσαν ούτε στην Ασία ούτε στην Ευρώπη του ΣΥΣΥΠΑ και έτσι βρισκόντουσαν εκτός ελέγχου όσων συμμετείχαν και των ρυθμιστικών αρχών και του δημοσίου. Τώρα 30 χρόνια μετά περίπου ρυθμίσεις που συζητούνται για αυτά τα τελευταία 30 χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών της δικής σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και της Επιτροπής του Κογκρέσου και παγκόσμια. 603 δολάρια. Για να σας δώσω ένα μέγεθος, αυτό σημαίνει 12 δολάρια για κάθε δολάριο που παράγεται παγκόσμια, οπουδήποτε σήμερα, είτε σε μια χώρα στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ ή στην Αφρική. Τώρα επιτέλους ήρθε η χρονική στιγμή πιστεύω να γίνουν μεταρρυθμίσεις και να γίνουν καινοτομίε σε αυτή την αγορά όπως και στην αγορά securities ή και στην αγορά on exchange, ε, futures markets. Πρέπει να είναι παγκόσμια και συνολική αυτή η προσέγγιση και να είναι επικοδομητική. Και έτσι λοιπόν όταν το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο όταν είχαμε του ηγέτες του G20 στο Pittsburgh συμφώνησαν όλα αυτά τα derivatives και όλα αυτά τα συμβόλαια να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στα χρηματιστήρια και να ελέγχονται και να στο τέλος του 2012 να βρίσκονται υπό εποπτεία. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε όλοι από κοινού σε αυτές τις προσπάθειες. Θεωρώ ότι η συνολική αυτή η ρυθμιστική μεταρρύθμιση πρέπει να καλύπτει όλους τους συναλλασσόμενους και όλα τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι τα προϊόντα σε σχέση με τα επιτόκια και τις ε, διακοιμάνσεις τους, ε, τα επιτόκια στις εξωτερικές αγορές, rate products, αλλά επίσης και αγαθά όπως ε, γεωργικά προϊόντα και οι, ε, πολλές φορές εξεταστήσα equity swaps και commodity swaps διαδικασία. Τρεις συνιστώσεις πρέπει εδώ να συμπεριλαμβάνονται που θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, ρύθμιση των ίδιων ε, των ε, συναλλασσομένων. Δεύτερον, διαφάνεια που πρέπει να αποκατασταθεί, ζητώντας να γίνονται με διαφανή τρόπο αυτές οι συναλλαγές. Και τρίτον, να υπάρχουν ε, κεντρικά ε, σώματα ή φορείς συμψηφισμού και ελέγχου. Πρώτον, για το πρώτο, για τους dealers, derivative dealers, είναι πολύ σημαντικό αυτές μεγάλες κεντρικές ε, ή μεγάλες, με συγχωρείτε, διεθνείς τράπεζες να βρίσκονται υπό εποπτεία όσον αφορά <clears throat> τα κεφάλαια και τις συναλλαγές τους αν δεν υπάρξει συμψηφιστική αρχή, αυτές οι transactions, αυτές οι συναλλαγές καταλήγουν σε μεγάλους κινδύνους. Αν δείτε παγκόσμια τι γίνεται, 14 μεγάλα θεσμικά παγκόσμια τέτοια κέντρα υπάρχουν που έχουν δεσπόζοντα ρόλο. 5-6 στη ΣΥΠΑ, 5-6 στην Ευρώπη και ένα ή στην Ασία. Αυτά τα 14-15 θεσμικά όργανα που είναι πολύ υπερβολικά μεγάλα και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να επιτρέψουν να τα αφήσουν να αποτύχουν, διασυνδέονται μέσω των derivative contracts. Και μέσω κεφαλαίου κινδύνου μπορούμε να μειώσουμε αυτούς τους κινδύνους. Επίσης οι dealers θα πρέπει να ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αξιόπιστες οι αρχές που θα διέπουν τις αγορές και να υπάρχουν ε, τρόποι τυποποίησης ε, των εγγράφων των συναλλαγών. Διάφορες λεπτομέρειες όσον αφορά συμβόλαια και παρόμοια πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι. Τέλος, όσον αφορά τους dealers είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πλήρη καταχώρηση των εγγράφων και συναλλαγών σε Μητρώα. Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ θα πρέπει να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση για να μπορούν να δουν τι γίνεται σε σχέση με τα συμβόλαια και τις συναλλαγές αυτών των dealers. Δεύτερον, πιστεύω πρέπει να προαρθεί η διαφάνεια σε αυτή την αγορά. Και σε αυτή τη διαφάνεια, αυτή η διαφάνεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο απαιτώντα ε, το να υπάρξει regulating, ρυθμιστική regulating platform κατά ιστερότερα ε, στο χρόνο όταν θα έρχεται θέματα και συμψηφισμού και κεφαλαίου κατά το καλοκαίρι και θα τα δούμε αυτά θα ήθελα να πω μόνο αυτή η διαφάνεια μπορεί να μειώσει κινδύνους ε, στο σύστημα διαφάνεια όσον αφορά τους ρυθμιστές δεν είναι επαρκή. Χρειαζόμαστε επίσης τη διαφάνεια για καλύτερες τιμέ και μικρότερου κινδύνους για όλους αυτέ αυτές τις συναλλαγές. Και έτσι νομίζω ότι αν θυμηθούμε για παράδειγμα τη ΣΥΠΑ είχαμε τον όρο τοξικά και ε, ομόλογα που δεν μπορούσαν να έχουν ε, συγκεκριμένη αξία. Και είχαμε τεράστιο όγκο δολαρίων που χρειάστηκε για να σωθούν ε, αυτές ε, οι τράπεζες, αυτά τα ιδρύματα να θυμηθούμε σε σχέση με την καταχώρηση εγγράφων και συναλλαγών. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά δεν επαρκεί αφέ αυτού. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε τι προσπάθειες στο Κογκρέσο που θα γίνουν και τι προσπάθειες από την Ευρωβουλή, ώστε να επιτευχθεί αυτό το διαφανέ πλαίσιο επιτέλου. Τρίτον, να αναφέρω τις over-the-counter derivatives και την ε, κατάληξή τους σε σώματα συμψηφισμού, υπηρεσίες συμψηφισμού. Προϊόν του τέλους του 19ου αιώνα και στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ έχουμε αυτή τη δράση ως μεσολαβητών μεταξύ συναλλασσομένων, διασφαλίζοντας ε, τα συμφέροντα φωτέρων σε αυτές τις συναλλαγές. Ένα clearing house για την επίτευξη αντιμετώπισης των δυσμενών περιόδων είτε πρόκειται για ύφεση και είτε αποτυχίες και χρεοκοπήσεις τραπεζών και είχαμε και τους πολέμους στο παρελθόν. Είχαμε λοιπόν τα χρήματα αυτά που μέσω των ε, ε, τραπεζών αυτών που ε, διαχειριζόντουσαν αυτά τα χρήματα όμως με αυτόν τον τρόπο ο καλύτερος τρόπος θα έπρεπε να δούμε ότι είναι η δυνατότητα συμψηφισμού και θα έπρεπε μια ρυθμιστική αρχή να επιληφθεί αυτού ώστε να έχουμε ένα καλύτερο διαφανέστερο πλαίσιο. Όσον αφορά το clearing houses, θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, επίτευξη υποχρεωτικής γεωγραφικής έδρας ε, για τέτοιου είδους συμψηφισμούς γιατί κάτι τέτοιο θα μείωνε την αποτελεσματικότητα της δράσης των κεφαλαίων. Το κυριότερο είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ρυθμιστές και εδώ ε, και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη θα έχουν σαφή και ανοιχτή πρόσβαση όσον αφορά τα στοιχεία των ε, Ιδρυμάτων Συμψηφισμού Συναλλαγών και ότι θα είναι αρκετά ισχυρά αυτά τα σώματα ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα από αυτά τα Ιδρύματα για τους φορολογουμένους μας. Τώρα, να πω δύο λόγια πέρα από αυτά τα τρία σημεία και να αναφερθώ περισσότερο σε κάποια άλλα θέματα που βρίσκονται και απασχολούν ε, τις ειδήσει και το, τους πολίτες. Για το swaps, ρύθμιση των dealers και μεγάλο διαφάνεια και έχοντας και αναγκαστική επιτήρηση εποπτεία μέσω clearing οδηγεί νομίζω σε αύξηση τη αξιοπιστία. όπως ε, και όσον αφορά την αγορά για τα επιτόκια αλλά αυτά όλα δεν θα υπαρκέσουν για τα swaps που έχουν ε, ιδιομορφίες. Οι ιδιομορφίες που τις κάνουν καμιά φορά να μοιάζουν σαν ασφαλιστικά συμβόλαια. Άλλες φορές να μοιάζουν σαν ε, ασφάλιση για παράδειγμα ομολόγων ή χρεογράφων πρόσθετα μέτρα που εξετάστηκαν στη ΣΥΠΑ και τα εξετάζουμε είναι ότι οι απαιτήσει κεφαλαίου για τις τράπεζες ε, που συναλλάσσονται θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι είναι παρόμοια ή έχουν ομοιότητες με ασφαλιστικά συμβόλαια, προϊόντα δηλαδή ασφαλιστικής αγοράς και όσοι εκδίδουν αυτά τα συμβόλαια εισπράττουν και ένα πριμ όπως και στα ασφαλιστικά συμβόλαια. Ξαφνικά όμως κάτι μπορεί να συμβεί, να χρεοκοπήσει η εταιρεία, να έχει προβλήματα και εμείς το λέμε αυτό ότι υπάρχει ένα πρόβλημα jump off, δηλαδή πρόβλημα κεφαλαίου. Κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσετε με ασφαλιστικά αποθέματα ή ε, κεφαλαιακά αποθέματα που διαφέρουν εκάστοτε. Το θέμα είναι αν το CDS, Credit Default Swaps, πρέπει να χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση αγορών. Και αυτό βρίσκεται υποσυζήτηση στην Ευρώπη σήμερα. Εμείς στη ΣΥΠΑ το εξετάσαμε και το είδαμε ως εξή. Είπαμε ότι οι αγορές έχουν κινδύνους μέσω κερδοσκόπων, μέσω δράσεων στην αγορά κεφαλαίου αν θέλετε να καλυφθείτε όσον αφορά τους κινδύνους για την αύξηση για παράδειγμα της τιμής ε, του πετρελαίου ένα τέτοιο swap μπορεί να είναι ή CDS μπορεί να είναι ένα μέσο. Υπάρχουν όμως και αρνητικές πτυχές. Αυτό που συστήσαμε στο Κογκρέσο είναι οι ρυθμιστικές αρχές, οι Securities Commission, να έχουν για παράδειγμα σαφείς εξουσίες να αντιμετωπίζουν χειραγωγημένες συναλλαγές και κερδοσκοπία ή κατάχρηση. Και αυτές θα είναι παρόμοιες με τις προστασίες που έχουμε στην αγορά συμβολέων ασφαλιστικών ή και futures συστήσαμε όμως κάτι παραπάνω. Συστήσαμε η Επιτροπή Ασφαλιών να έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα για το position limits, τα όρια θέσεων, αυτό, ε, τα όρια συναλλαγών. Αυτό θα περιόριζε κάποια συναλλαγέ. Αν ένα λοιπόν θέμα η μια εταιρεία αρχίζει να αγοράζει κάποια bonds ή securities derivatives και CDS προσθέτονται συσσωρευτικά, τότε θα μπορούσαν να έχουν ένα όριο οι ρυθμιστικές αρχές που θα θέτουν για τέτοιου είδους σορευτικά συναλλαγές. Επίσης και όσον αφορά το, την πρόταση που θα υποβληθεί από πλευρά ΙΠΑ θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί από πλευρά της Γερουσίας, Σένετ. Υπάρχει και κάποιο θέμα για κάποιες εξαιρέσεις. Μιλήσαμε με πολλές εταιρείε και πολλούς ε, ε, τραπεζίτες και είπαν καλό είναι να προχωρήσετε σε αυτή τη μεταρρύθμιση αλλά μπορούμε εμείς να εξαιρεθούμε. Γίνεται αυτό και στην Ευρώπη εδώ επίσης. Σας ζητάνε τέτοιες εξαιρέσεις. Ε, όμως συμβαίνει στη ΣΥΠΑ βλέπετε. Και πρέπει όμως πιστεύω να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα συμβόλαια στην κεντρική αυτή αρχή ρύθμισης και συμψηφισμών. Και υπάρχουν εδώ οι απαιτήσει για εξαιρέσεις και εδώ υπάρχουν ανησυχίες για αύξηση ε, κόστους, ε, ε, αύξηση κεφαλαίου. Τώρα, δεν είναι το θέμα των derivative contracts, αλλά είναι το αίτημα αυτών των... Αν αφήσουμε όμως γενικά αυτές τις εξαιρέσεις, αυτό υπονομεύει και περιορίζει πολλές από τις μεταρρυθμίσεις. Και είδαμε το 2008, όταν δεν είχαμε ότι όταν είχαμε τους φορολογουμένους ε, που βρισκόντουσαν, ε, αναγκάστηκαν να τροφοδοτήσουν με χρήματα τους, ε, τις τράπεζες. Είναι λοιπόν τέτοιου είδους αυτά τα θέματα που θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Και προτείνω να δούμε το πώς γίνονται αυτά τα πράγματα σε σχέση με τις σε σχέση με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία. Οι συναλλαγές μεταξύ dealers και non-financial corporations Έχουμε δηλαδή ε, παροχή υπηρεσιών, λιανικό εμπόριο, συνολικά 9% όλων των συναλλαγών. 57% των συναλλαγών μεταξύ των τήρεση και άλλων ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι αυτό. Και είναι σημαντικό αυτές οι συναλλαγές να ενταχθούν μεταξύ μεγάλων τραπεζών και ασφαλιστικών ε, εταιριών ή και hedge bonds γιατί να αφήναμε αυτές τις συναλλαγές μεταξύ hedge funds και τραπεζών ή hedge bonds εκτός αυτών των ρυθμίσεων. Υπάρχει το θέμα της εξαίρεσης συναλλαγών μεταξύ τραπεζών για παράδειγμα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν ήθελα να επιλέξω μόνο μία από αυτές τις ε, δραστηριότητες. Σίγουρα μπορούν να εξεταστούν και άλλες. Αλλά ας αναφέρω κάτι τώρα προτού ολοκληρώσω σε σχέση με τα παράγωγα. Και όπως γνωρίζετε αυτό έχει αναφερθεί και σε σχέση με ειδήσει πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά οι διάφορες χώρες ως μέσο. Έχουμε εδώ σε σχέση με τα παράγωγα όσον αφορά το θέμα του χρέους της Ελλάδας για παράδειγμα και τεκτενόμενα και αλλού σήμερα αυτή τη συζήτηση. Τα παράγωγα διαδραμάτισαν ένα ρόλο σε αυτό, κάποιο ρόλο και το είδαμε και στις ειδήσει. Δημοσιεύματα λένε ότι κάποιες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει συμβόλαια derivatives όσον αφορά τις off-market transactions. Δηλαδή εκεί όπου έχουμε μέσα σε ένα παράγωγο και ένα δάνειο το οποίο εντάσσεται εκεί το derivative, το παράγωγο, έχει κάλυψη κινδύνου. Όπως, όμως τουλάχιστον μία χώρα, ε, η Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια, ένα δις είχε εντάξει μέσα σε παράγωγα. Εγώ δούλεψα στη Wall Street, στο χρηματιστήριο, πάνω από 18 χρόνια και ξέρω αυτά τα πράγματα και όποιο θέλει διμερώς να τα συζητήσουμε μετά την ακρόαση είμαι στη διάθεσή του. Σε σχέση με τέτοιου είδου ε, ε, συναλλαγέ θα μπορούσαν να οδηγηθούν στην κεντρική ρυθμιστική αρχή συμψηφισμού και όταν θα γίνει αυτό δεν θα μπορεί κανεί να ε, έχει την επέκταση ενό τέτοιου δανείου ενό δι σε παράγωγα γιατί θα υπάρχει και όριο. Αν θα ήθελε κανείς διμερός να το δει, νομίζω οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν σαφή εντολή για τη ρύθμιση αυτών των αγορών. Να θέσουν τόσο υψηλά τις προδιαγραφές ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου είδους συναλλαγές. Είναι ένα απλό παράδειγμα. Να υπενθυμίσω γιατί χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την Πρόεδρο με αυτή την παρατήρησή μου. Ολοκληρώνω έτσι. Η διεθνή συντονιστική προσπάθεια λειτουργεί σε ένα σημαντικό αξιοπρόσεκτο βαθμό Βρισκόμαστε στην ίδια πορεία και διαδρομή παρότι έχουμε διαφορετικά, ε, διαφορετικές παραδόσεις. Αντιμετωπίζουμε όμως τα ίδια προβλήματα θέλοντας να διασφαλίσουμε μικρότερους κινδύνους ε, για τους πολίτες μας, διασφαλίζοντας επίσης και την αύξηση της διαφάνειας είναι πολύ περίπλοκο αυτό το πλαίσιο, αλλά συνεργαζόμενοι από κοινού μπορούμε να καταλήξουμε, ελπίζουμε, κατά τα τέλη του 2010 να τα καταφέρουμε, ώστε να μην, θέτονται, τίθενται μεγάλα προβλήματα από τι ε, διεθνεί τράπεζε όπω μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σα για απάντηση ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνεισφορά σας. Ήδη έχουν ζητήσει το λόγο αρκετοί. Ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να ρωτάμε μία ερώτηση κάθε φορά και αν δούμε ότι δεν έχουμε χρόνο μετά τις ακούμε αναομάδες. Ποιος άλλος? Podimata, Catherine Styler, Sven Giegold. Anybody else? Alos. Any advance on Vicky Ford? Um, um, maybe we better take you two at a time. Ας ξεκινήσουμε τότε με δύο ερωτήσεις κάθε φορά. Κλείσει. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε και για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μία ευρία και απλή ερώτηση. Είπατε ότι το εμπόριο δεν γνωρίζει σύνορα. Τώρα όμως με αυτή την κρίση που την αντιμετωπίζει και η ευρωπαϊκή και η αμερικανική πλευρά. Προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας ό,τι μπορούμε. Μήπως όμως θα ήταν καλύτερα να έχουμε μια πιο δομημένη διαδικασία διασύνδεσης των διαδικασιών μας. Γιατί και των δύο πλευρών οι διαδικασίες είναι περίπλοκες. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο αν έλθουμε σε επαφή προκειμένου να μην δημιουργηθούν ανισορροπίες μεταξύ των ρυθμιστικών μέτρων που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από την πλευρά σας τι είδους ε, δομικές διασυνδέσεις θα προτείνατε προκειμένου να έχουμε ένα εναρμονισμένο συναφές ρυθμιστικό πλαίσιο στα πλαίσια των διαφόρων διεθνών συμφωνιών, ενδεχομένως ε, διεθνών επιτροπών. Θυμηθείτε το αυτό και περνάμε στον Ούντο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών για την επίσκεψή σας και σας ευχαριστούμε επίσης για την φρέσκια και ανοιχτή προσέγγισή σας. Αναφερθήκατε σε ορισμένες ομοιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής. Μία ομοιότητα είναι ότι όλοι θεωρούν ότι πρέπει να ρυθμιστούν όλοι οι φορείς εκτός από τους δικούς μας. Εκτός από εμάς. Κάτι άλλο. Από τη μία πλευρά γίνονται πολλές συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις, αλλά από την άλλη όταν ερχόμαστε σε συγκεκριμένα θέματα τα πράγματα μπερδεύονται. Ένα ερώτημα λοιπόν. Πώς πιστεύετε ότι θα μοιάζει το πακέτο μετά την εμπειρία της Γερουσίας. Δεύτερον, κατά τη γνώμη σας, ο ρυθμιστικός οργανισμός θα είναι μία αρχή που θα εφαρμόζει πολύ αυστηρές υποχρεώσεις ή θα πρέπει να είναι πολύ ευέλικτος όσον αφορά τους διαφορετικούς φορείς τις διαφορετικές χρονικές στιγμές ή άλλες ε, συνθήκες προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης. Κάτι άλλο. Στην Ευρώπη μιλήσατε για τις ε, αγορές αγαθών. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ρύθμιση αν αποκλειστούν οι αγορές αγαθών. Ευχαριστώ για τις πολύ καλές ερωτήσεις. Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ευρώπη σήμερα. Βεβαίως με ρωτήσατε αν δεν κάνω λάθος και πώς θα συνεχιστεί η συνεργασία. Επί της ουσίας νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν τα ίδια πράγματα υψηλά κεφάλαια για τα προϊόντα που έχουν ε, συγκεκριμένη χρήση. Τι μπορεί να γίνει. Καταρχάς, η νομοθεσία στην Αμερική που σέβεστε και εσύ δεν επιτρέπει σε μία αρχή να βλέπει τα στοιχεία άλλης. Βεβαίως, αυτά τα στοιχεία μπορεί να ενδιαφέρουν και τις άλλες πλευρές γιατί οι 14 μεθυστικές αρχές θα έχουν διεθνή εμβέλεια και επομένως θα χρειάζονται οι ρυθμιστικές αρχές στο Λονδίνο ή στο Παρίσι αυτά τα στοιχεία και είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρχει ανταλλαγή τους. Περνάω στην επόμενη ερώτηση. Ναι, θα πρέπει να έχουν περιθώρια ευελιξίας οι ρυθμιστικές αρχές. Πρέπει να υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις που να απαιτούν τη χρήση του κεντρικού οργανισμού συμφισισμού. Θα έπρεπε να υπάρχουν λοιπόν σαφείς προϋποθέσεις για το ποιες συναλλαγές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Όσον αφορά τη γερουσία, εγώ ως ε, αιώνιος αισιόδοξο θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε ένα νομοσχέδιο που θα ψηφίσει ο πρόεδρός μας, αλλά ενδεχομένως στο τέλος του έτους. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, θα υπάρξει ένα νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση που θα υπογραφεί φέτος. Μας ενδιαφέρουν θέματα που έχουν να κάνουν με τους χρηματιστές, τους dealers και τα υψηλά κεφάλαια και θεωρώ ότι υπάρχει σαφή συνένεση προκειμένου να απαιτούνται υψηλές προκαταβολές και επίσης φαίνεται να υπάρχει συνένεση και για το θέμα της κεντρικής αρχής συμψηφισμού, αλλά ζητούνται πολλές εξαιρέσεις. Εγώ είμαι κατά, όμως βεβαίως ε, ο επιχειρηματικός κόσμος ε, επιμένει επί του θέματος αυτούς. Δεν γνωρίζω πού θα καταλήξουμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να καλύψουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το τελευταίο θέμα, όσον αφορά την ε, διαφάνεια στην Βουλή των Αντιπροσώπων για να πω κάτι που ίσως προκαλέσει. Η Wall Street είναι αλλεργική στο θέμα αυτό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι παίκτες ε, του χρηματοπιστωτικού παιχνιδιού δεν θέλουν να δοθεί αυτού του είδους η ενημέρωση στο κοινό και όσον αφορά τα παράγωγα. Πρέπει να καλυφθούν τα παράγωγα. Είχαμε ξεκινήσει την δεκαετία του 20. Τότε όλα συμπεριλαμβάνονταν στο χρηματιστήριο. Δεν μπορούσαν να γίνουν έξω χρηματιστηριακές πράξεις. Σήμερα, 80-90 χρόνια μετά, έχουμε πολλά έξω αγαθά όπως ε, τα σιτηρά ή το πετρέλαιο. Και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος προστασίας του κοινού, ειδικά εφόσον πρόκειται για προϊόντα για τα οποία έχουμε πεπερασμένα αποθέματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε εκμετάλλευση και στρεβλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Βόλφ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε τους ε, στόχους σας για μεγαλύτερη διαφάνεια, μείωση των κινδύνων και ελαχιστοποίηση των ε, δυνατοτήτων ε, στρέβλωσης. Είχαμε μία συνάντηση με την Πόνη Φρανκ ε, και είχε συζητηθεί και το θέμα των κεντρικών οργανισμών συμψηφισμού και είχε αντιδράσει αρκετά αρνητικά. Είχε πει ότι ισοδυναμούσε σχεδόν με κηρύξη πολέμου τότε δεν του είχε αρέσει καθόλου λοιπόν αυτή η ιδέα γιατί φοβόταν ότι οι επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις Ηνωμένε Πολιτείε θα μετανάστευαν προς την Ευρώπη. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω, αν έχει όντως αλλάξει άποψη, τι τον έκανε να αλλάξει άποψη. Δεύτερο θέμα. Καταστήσατε σαφές ότι προκειμένου να έχουμε διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών αγορών θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνής προσέγγιση. Διαφορετικά θα δημιουργηθούν ανταγωνισμοί και δυνατότητες επιλογής ανταγωνιστικών διαιτησιών κτλ. Κάτι όχι καλό. Τώρα, αν σκεφτεί τον όγκο 600 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όχι μόνο χρειάζεται καλή ρύθμιση, αλλά πρέπει να μειωθεί και ο όγκος, γιατί μεγάλο ποσοστό αυτό του συναλλαγών είναι καθαρά κερδοσκοπικές. Δεν έχει καμία οικονομική συνεισφορά. Όταν έχω αυτοκίνητο, θέλω να έχω ασφάλιση έναντι ατυχημάτων. Αν όμως δεν έχω αυτοκίνητο δεν χρειάζομαι ασφάλιση. Γιατί λοιπόν να πρέπει να έχουμε ασφάλιση ανταλλαγής κινδύνων αν δεν έχουν κάποιους κινδύνους. Για παράδειγμα, αν δεν έχουν ελληνικά ομολογά, γιατί να χρειάζονται τέτοιου είδους ασφάλιση. Θα έπρεπε αυτού του είδους οι πράξεις να εξαφανιστούν κατά τη γνώμη μου. Και περνάω στο θέμα των κεντρικών οργανισμών συμψηφισμού. Μήπως θα έπρεπε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που ελέγχουν αυτό το εμπόριο δεν θα είναι εταίροι αυτών των κεντρικών οργανισμών συμψηφισμού. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε νομίζω ότι κινδυνεύει το όλο εγχείρημα. Ευχαριστώ και το λόγο έχει και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά με ενδιαφέρει πολύ το θέμα και συχνά γίνομαι αρκετά έντονη. Κοιτάξτε, στην δική μου περιοχή που είναι μάλλον αγροτική περιοχή υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν μικρά περιθώρια κέρδου. Αν λοιπόν δεν μπορούν να έχουν κάποια αντιστάθμιση του κινδύνου τότε μπορεί να καταλήξουν σε χρεοκοπία. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να κάνουν ε, συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνων για όλα, για οτιδήποτε, επειδή έχουν μικρά περιθώρια ε, κέρδους. Αν για αυτές τις επιχειρήσεις υπάρξει εξαίρεση, θα ήθελα να γνωρίζω πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτό. Και επίσης να πω, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά μεταξύ του να πωλείται ένα παράγωγο για hedging, για αντιστάθμιση κινδύνου ή για παροχή overdraft. Τι σημασία έχει το τι είδους εργαλείο χρησιμοποιούμε αν ουσιαστικά η τράπεζα το πολύ για τον ίδιο σκοπό. Νομίζω ότι οι τράπεζες εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία και δεν θα έπρεπε να αλλάξουμε τις σχέσεις πελάτη-τράπεζας κατά αυτόν τον τρόπο. Ένα άλλο θέμα, αυτό της ε, διαλειτουργικότητας ε, των συμβάσεων των ε, κεντρικών οργανισμών συμψηφίσμου. Μήπως αντί να έχουμε μεμονωμένους τέτοιους οργανισμούς συμψηφισμού που δεν θα επιτρέπουν στους πελάτες να μεταβαίνουν από τη μία πλατφόρμα στην άλλη Μήπως θα έπρεπε να έχουμε κάποια διαφορετική διαλειτουργικότητα, κάτι που θα βοηθούσε τους πελάτες. Και κλείνω με κάτι αρκετά προκλητικό. Τι κάνουμε στο μέλλον, γιατί να σταματήσουμε στα παράγωγα, γιατί να μην ζητήσουμε διαφάνεια για όλες τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, όχι μόνο τα παράγωγα. Φοβάμαι ότι επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα σημείο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και μπρος η Αμερική εξαιρετικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αν γίνεται. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο και θα καταλήξω για την κεντρική συμψηφιστική εταιρεία. Για τον τελικό χρήστη end νομίζω θα υπάρχει μεγάλη συμφωνία σε σχέση με το μέλος ε, Ευρωβουλευτή που έθεσε την ερώτηση ότι οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να καλύπτουν τους κινδύνους των συναλλαγών τους και εμείς θέλουμε να προαγάγουμε συναλλαγές, οικονομικές συναλλαγές αλλά να μειωθούν οι κίνδυνοι από πλευρά συστήματος. Αν είναι μια τέτοιου είδου συναλλαγή στάνταρτα με μικρότερου τέτοιου κινδύνου και που θα καταλήγει στο συμψηφιστικό όργανο αλλά για το τελικό που αναφέρατε πρόκειται για ένα overdraft, συμφωνώ με αυτό. Αν εξαιρεθεί από τους συμψηφιστές αφήνεται μεγαλύτερος κίνδυνος, κάπως μεγαλύτερος κίνδυνο στο σύστημα και για τους μικρούς εμπόρους ε, που συναλλάσσονται όσον αφορά για παράδειγμα με τα σιτηρά θα ήταν σημαντικό να μην εξαιρέσουμε τις ε, χρηματικές συναλλαγές ε, με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά εκτός πλαισίου. Ακόμα και αυτός ο έμπορος σιτηρών βαρύνεται έχουμε charge credit το οποίο καλείται να πληρώσει. Και αν υπάρχει overdraft πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα καλύπτει τέτοιου είδους ε, δράσεις ε, ως εγγύηση. Εδώ βρισκόμαστε. Στη ΣΥΠΑ θα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ε, τελικών χρηστών και αυτό αναφέρθηκε και σε σχέση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αλλά περίπου θα έλεγα 8-9% της αγοράς, όχι 60-65% της αγοράς. Τρεις ερωτήσεις βρισκόντουσαν στην παρέμβασή σας, ε, στις παρεμβάσεις σας για τις ε, ε ρυθμιστικές ε, συμψηφιστικές αρχές. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει open access, να υπάρχει ανοιχτή προσπελασιμότητα, πρόσβαση σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές δεν είναι αυστηρά διαλειτουργικότητα. Σημαίνει ότι σε σχέση με μια τέτοια συμψηφιστική αρχή θα πρέπει να εντάσσονται οποιασδήποτε τέτοιε συναλλαγέ. Και με αυτή την επιτήρηση θα έχουμε προαγωγή του ανταγωνισμού. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία ισχύουν με τα μελλοντικά παράγωγα. Δεν είναι το ίδιο. Επίση, πιστεύουμε ότι οι συμψηφιστικέ αρχέ πρέπει να έχουν open governance, ανοιχτή διακυβέρνηση. Και αυτό αφορά και την ερώτηση αν θα πρέπει να περιοριστεί το θέμα ιδιοκτησία ή όχι. Το πιο σημαντικό όμω είναι οι ρυθμιστές να μπορούν να υποπτεύουν την διαχείριση και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα συγκρούσεως αρμοδιοτήτων άσχετα από το ποια θα είναι η ιδιοκτησία, αν θα είναι μία ή αν θα είναι κοινή ε, συμμεριζόμενη, θα πρέπει να εποπτεύονται από τις συμψηφιστικές αρχές. Ο πρόεδρος ε, Φρανκ πέρασε ένα νομοθέτημα ιστορική σημασίας από την Επιτροπή μας πέρυσι και έτσι όποιε και να ήταν οι σκέψεις του πριν από 1,5 χρόνο θα έλεγα ότι είναι πλέον σαφέ ότι ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα πέρασε και εγκρίθηκε μέσα από, μέσα από την Επιτροπή αυτή. Και έτσι, σε σχέση με την ε, τελική εξαίρεση για κάποιους χρήστες, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει εντολή σε σχέση με ένα συμψηφιστικό όργανο να μην δεσμεύονται αυτά τα όργανα με κάποια έδρα, να μπορούν να έχουν την έδρα τους ε, όπου ε, χρειάζεται, όπου είναι αναγκαίο. Και για το CDS, Credit Default Swaps, Νομίζω ότι υπάρχουν ε, μοναδικές ε, ιδιομορφίες για τα CDS, ιδιαίτερα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ε, χειραγωγήσει κάποιος μια αγορά ή ίσως το χρέος και μια χώρας ή το θέμα του χρέους μιας εταιρείας. Το θέμα αυτό που όπως το προσεγγίζουμε εμείς στη ΣΥΠΑ, που δεν είναι η μόνη σωστή προσέγγιση, αλλά είναι μία προσέγγιση, θέλουμε οι ρυθμιστικές αρχές να έχουν σαφή πρόσβαση, ώστε να εποπτεύουν και να επιβάλλουν τους κανόνες ε, και τη συμμόρφωση με αυτούς και να υπάρχει και όριο σε σχέση με το τελικό επίπεδο συναλλαγών. Εγώ δεν ξέρω ευθύ εξ αρχή να πω πώ μηχανικά θα μπορούσε κάτι τέτοιο ε, εκ να πούμε ότι αυτόματα θα λειτουργούσε σεβόμαστε ότι μια οποιαδήποτε απαγόρευση συλλήβδη για την οικονομία όχι μόνο είναι δύσκολο να υποπτεύεται αλλά προτού το κάνουμε και την υιοθετήσουμε μια και είναι σημαντικό εμπόδιο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνετοί. Πρέπει όμως εδώ να προστατευτεί η αγορά κατά, κατά χειραγώγησης και στρεβλώσεων και ε, κατάχρησης και γι' αυτό λοιπόν προ, τίνεται μια τέτοια δράση. Νομίζω ότι με την απάντησή μου κάλυψα σε σχέση με το position limits, τα όρια αυτά. Αυτά αναφέρονται πάντα σε σχέση με, τα, τι, με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάποιο δόγμα ή έχει καθοριστεί ευθύ εξ αρχή. Έτσι δεν είναι. Και το άλλο, στο οποίο ίσω δεν απαντήσατε πλήρω για τα 603 και πόσα από αυτά είναι κερδοσκοπία ή όχι. Ναι, σα ευχαριστώ που μου το υπενθυμίσατε. Και επίση βλέπω ότι υπάρχει και ένα θέμα για το μέχρι πού πρέπει να φτάνει η διαφάνεια. Για το position limits, τα όρια συναλλαγών και σε σχέση με το 1930 όσα συνέβησαν στον τομέα των γεωργικών αγαθών και των αγαθών. Με βάση κάποιο τύπο υπολογισμού είπαμε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πολυμορφία των ε, εμπλεκομένων. Να υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί που θα ισχύουν για τους εμπλεκόμενους και όλοι να τους γνωρίζουν τα όρια και τα, ε, τους κανονισμούς. Να υπάρχει ε, ένα, τέτοιο σώμα κανονισμών. Αλλά και υπάρχει εδώ κατ' εντολήν ε, κατανάθεση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές αυτό το θέμα για να το ρυθμίσουν οι ίδιοι. Για τα 603 δεν ξέρω ποιο είναι το ακριβές ποσό της ε, κερδοσκοπίας και κανείς δεν νομίζω να το ξέρει. Ε, είναι μια πρόκληση αυτή. Είναι ένας, θα το έλεγα, περιόριστος τομέας αυτή η αγορά. Πρέπει πραγματικά να εισαγάγουμε το θέμα της διαφάνειας ε, σε αυτούς τους εμπλεκόμενους σε αυτές τις αγορές για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Υπάρχει εδώ ένας ρόλος για αυτούς τους κερδοσκόπους που συναντούν τους hedges, εκείνους που δρούν με κεφάλαια αμοιβαίου κινδύνου σε αυτές τις αγορές. Αλλά ξέρουμε το ακριβές ποσοστό. Η αγορά παραγόγων σήμερα έχει ε, σημαντικές επιπτώσεις ε, και υποβάλλεται σε κάποιες διαδικασίες συγκεκριμένες. Όλες αυτές οι εταιρείες ε, και όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι που προαναφέρθηκαν. Είναι όμως και πολύ υπάρχει μεγάλη δυνατότητα μέσω των κομπιούτερς, των υπολογιστών και του συστήματος στο διαδίκτυο. Έχουμε και το θέμα των securities markets και future markets αυτό στις είπα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι το επόμενο κέριο βήμα που πρέπει να γίνει. Αν μπορεί κανείς να το ε, συστήσει αυτό και για άλλες αγορές, σίγουρα. Αλλά είναι νομίζω ένα κύριο, κύριο στοιχείο στην κρίση αυτή που πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτή τη δράση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλίν και μετά Πεβάνς, παρακαλώ. Μια φιλοσοφική θα έλεγα στοχαστική ερώτηση. Είπατε ότι συνεχίζεται αυτή η ρυθμιστική προσπάθεια. Υπάρχει όμως μεγάλη επιρροή από το χρηματιστήριο στη ΣΥΠΑ, του Wall Street και ότι είσαστε ε, αισιόδοξο. όμως ε, εδώ σε σχέση με τον, ε, την αισιοδοξία αυτή ίσως δεν θα μπορούσα να την συμμεριστώ κι εγώ. <clears throat> Έχουμε 344 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με λομπιίστες, έχουμε δώρα τα οποία δίνονται σε σχέση με μέλη επιτροπών. Δεν είμαι τόσο οπτιμίστρια. Σε σχέση με τα CDS Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει απαγόρευση για τέτοιου είδους ε, ε, CDS συναλλαγές ή όχι. Και λαμβάνοντας υπόψη ε, το μικρό αριθμό funds που εμπλέκονται, γιατί είπατε ότι υπάρχουν κίνδυνοι σύγκρουση συμφερόντων πιο πριν, πιστεύετε ότι είναι εύθετο και σκόπιμο όταν έχει δεσπόζοντα ρόλο από μια, ε, η αγορά από πλευράς μικρού αριθμού συναλλασσομένων και στο CDS θα, θέλατε να σχολιάζατε το θέμα των ερευνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αυτόν τον τομέα ή όχι. Σας ευχαριστώ. Πολύ πονηρή ερώτηση. Να θέσω και εγώ τη διαρώτηση με την Αρλίνη σχετικά με την σημασία των χρημάτων που δαπανά, ο χρηματοοικονομικός, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος για να με, έχω ένα άλλο στοιχείο. Εγώ 400 δις ευαισθητούστε η διαφορά δεν είναι και μεγάλο, της έχει τη δική του αντίληψη περί δημοκρατίας. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε όμως κάποια φάκελοι που υπάρχουν στο Κογκρέσο και να εξεταστεί και η πραγματικότητα αυτών των στοιχείων. Τώρα έχω τρεις ερωτήσεις. Η μία έχει ως εξής. Εδώ στην Ευρώπη από τότε που ε, δημιουργήσαμε ένα σύστημα ε, διάσωση των τραπεζών δεν πετύχαμε και πάρα πολλά όπως και σε εξάρτου αλλά κάναμε κάτι προχωρήσαμε σε ό,τι αφορά το πακέτο επιτήρηση όταν ρίχνουμε μια ματιά στην κατάσταση όπως αυτή επικρατεί δηλαδή στην Αμερική ε, δεν ξεκινάμε από το ίδιο σημείο κίνηση. υπάρχει το λεγόμενο spaghetti ball πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την απορρόφηση του spaghetti ball δεν θα ήθελα να κάνω κάποια σύγκριση διατροφ, διατροφής, αλλά και μια δεύτερη ερώτηση. Πώς συλλογείται τις τελευταίες προτάσεις ε, του Πρόεδρου Ομπάμα σχετικά με τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του G20. Νομίζω πως η ατζέντα του G20 ε, ετοιμάστηκε σε στενή συνεργασία από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και όταν μιλούσαμε για μια ενίσχυση των ιδίων ε, κεφαλαίων αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη ούτε για το Υπουργείο Οικονομικών ούτε για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αυτό όμως ε, φαίνεται ότι δεν είναι και το βασικό σημείο και το ονομαζόμενο πακέτο Volcker αποτελεί μια στροφή 180 μοίρων σε σχέση με τα συμπεράσματα του G27. Τι σημαίνει ότι δεν το είχατε σκεφτεί προηγούμενα, θεωρήσατε ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην κοινή ατζέντα κάτι τέτοιο και τρίτη ερώτηση προκειμένου για τα ΣΕΝΤΕΣ συμβάσει ανταλλαγή κινδύνου αθέτηση. Δέχεστε την. Και όχι μόνο δέχεστε, αλλά δεν θεωρείτε ότι είναι σκόπιμη, απαραίτητη, αναγκαία. Να υπάρχει λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως και στην ζώνη Ρο ένα γραφείο ε, συμψηφισμού των ΣΕΡΕΣ στην περίπτωση της Ελλάδας πραγματικά βρεθήκαμε κάπως ε, ανέτοιμοι διότι υπήρχε ένα ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία των ΣΕΝΤΕΣ και ήσασταν η μοναδική αρχή που είχατε τις προφορίες σχετικά με την πραγματικότητα του πώς λειτουργεί αυτή η αγορά. Κάτω ποιες προϋποθέσεις λοιπόν δέχεστε να χορηγείτε προφορίες ανάλογα με τις κινήσεις που έγιναν στα ΣΕΝΤΕΣ και που και πώς βλέπετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ενός, μιας υπηρεσίας μου στην Ευρώπη και κατά ποιε προϋποθέσεις δέχεστε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη στις αγορές των ΣΕΝΤΕΣ. Ευχαριστώ. Um, Θα έλεγα και τα δύο μέλη ευρωβουλευτές ε, και σε σχέση και με τη φιλοσοφική μορφή ερώτηση που τέθηκε εγώ ίσω από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο. Είναι οι κόρε μου εδώ, μπορούν να σας το πούν ίσω καλύτερα αυτό. Ζούμε όμω σε αυτέ τι ε, δημοκρατικές χώρες και ο κάθε μπορεί να ε, έχει τα επιχειρήματά του, ακόμα και το χρηματιστήριο στη ΣΥΠΑ, η Wall Street. Πρόκειται για το ποιος έκανε το αυγό η κότα ή το αυγό έκανε την κότα. Δεν μπορείτε να λέτε ότι έχετε άμεση πρόσβαση. Ε, από τη μία πλευρά υπάρχει η τράπεζα και από την άλλη υπάρχει το... Έχετε αμεση προσβαση απο τη μια πλευρα υπαρχει η τραπεζα δίκιο σε αυτά που λέτε κύριε Ευρωβουλευτά. Η Wall Street έχει πάρα πολλά επιχειρήματα ε, που χρησιμοποιεί και πολλές φορές ε, οι υπόλοιποι Main Street ε, δεν έχουν. Εμείς όμως υποστηρίζουμε αυτό που η CFTC λέει και από πλευρά ε, κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρξουν αυτές οι ρυθμίσεις. Απέτυχε το χρηματιστήριο, το η Wall Street, όχι μόνο στη ΣΥΠΑ αλλά και παγκόσμια έναντι των πολιτών. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ καλή κατανόηση αυτών των πραγμάτων στο Κογκρέσο στη ΣΥΠΑ. Μπορεί να μην πετυχαίνουμε όλα αυτά τα οποία ζητά και ζήτησε ο Πρόεδρος ίσως και αυτά που εγώ ζητώ. Εντάξει, όμως, τούτου λεχθέντος πιστεύω ότι μεγάλο βήμα προς τα εμπρός μπορεί να επιτευχθεί, μειώνοντας τους κινδύνους σε αυτές τις αγορές παραγόγων στις συναλλαγές. Και πάλι όμως θα με θεωρήσετε ε, αισιόδοξο. Σε σχέση με τις λεπτομέρειες για τα CDS, Credit Default Swaps, νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα πολύ ισχυρό πακέτο δέσμη μέτρων ρύθμιση των συναλλασσομένων. Αυτέ οι συναλλαγέ όχι μόνο πρέπει να καταλήγουν σε κεντρικέ συμψηφιστικέ αρχέ, αλλά πρέπει να είναι και διαφανεί. Πρέπει το κοινό να έχει προσπελασιμότητα πρόσβαση ώστε να είναι διαφανέ το πλαίσιο. Και επίση πρέπει να υπάρχει επόπτευση, ε, επιτήρηση ώστε να υπάρχει συμμόρφωση κανονισμών. Και αυτό ίσω διαφοροποιεί ε, το αν ε, θέλουμε να υπάρξει απαγόρευση ή όχι για το CDS. Δεν ξέρω πως κάτι τέτοιο απαγόρευση θα μπορούσε να λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, παρέμβαση εκτός μικροφώνου, μίλησα ίσως ε, υπερβολικά σύντομα, αλλά ακόμα και η γυμνή, το Naked CDS, Credit Default Swaps. Και εδώ, σε σχέση με μια παρέμβαση που έγινε, τουλάχιστον εμείς στην έρευνά μας, εδώ και με την αυτιλία πολύ καιρό παλιότερα, ότι ασφάλεια μπορεί να γίνεται μόνο σε σχέση με ένα πλοίο και ένα φορτίο. Ξεκινά αυτό από ήδη αιώνε πριν από την ε, Μεγάλη Βρετανία. Έχει ζητηθεί ο ρόλο των κερδοσκόπων στι αγορέ και στι συναλλαγέ και από την περίοδο του, της βασιλείας του βασιλέως Γεωργίου του Δευτέρου ή ακόμα και νωρίτερα. Όμως οι κερδοσκόποι στις αγορές υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στη ΣΥΠΑ είναι να παίρνουμε αυτές τις πληροφορίες, να διατίθενται οι πληροφορίες, όλες οι ρυθμιστικές αρχές να τις έχουν, να αποκατασταθεί η διαφάνεια προς το συμφέρον των πολιτών, του κοινού και να έχουν οι ρυθμιστικές αρχές να αντιμετωπίσουν αυτές τις συναλλαγές ε, με ρυθμιστικές διατάξεις και ανώτατα όρια για τις συναλλαγές. Τώρα, ίσως σε σχέση τώρα με τις άλλες παρεμβάσεις που έγιναν, ερωτήσεις σας θέλω να είμαστε σίγουροι ότι αυτές θα μπορέσουν να απαντηθούν αυτές οι άλλες. Φυσικά δεν μπορώ να σχολιάσω για τις έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης της ΕΠΑ. Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό ως παρέμβαση. Σύγκρουση αρμοδιοτήτων τώρα που έγινε. Λέγεται στον ομιλητή εκτός μικροφώνου κάτι, δεν το ακούμε, οι διερμηνείς. Αν, να, αν δεν μπορεί να απαντηθεί, να ξαναρωτηθεί η ερώτηση αυτή η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν αν θεωρείτε εσείς προσωπικά ότι υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων εδώ σε σχέση με τραπεζικό όργανο, ε, τράπεζα που, ε, μείζωνα τράπεζα που εργάζεται σε σχέση με αυτό τον τομέα, δραστηριοποιείται εκεί. Συγγνώμη, λέει ο μιλητή. Νομίζω ότι η επικέντρωση στην ε, χρηματοοικονομική κοινότητα, είτε βρίσκεται αυτή στη Wall Street, στη ΣΥΠΑ, είτε εδώ στην Ευρώπη, είναι κάτι που ανησυχεί έντονα. Αυτή η συμπίκνωση δραστηριοτήτων, η επικέντρωση αρμοδιοτήτων, οδηγεί πρώτον σε μεγάλο κίνδυνο που έχουν οι φορολογούμενοι, που πρέπει εκείνοι, αν υπάρξει κίνδυνος, να καλύψουν τις ζημιές όταν έχουμε ε, διασυνδεόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αυτό είναι ένα κίνδυνο. Άλλο κίνδυνο αυτού του πριτανεύοντο ε, ρόλου είναι ότι η διαμόρφωση των ε, τιμών του πλαισίου τιμών δεν είναι τόσο αποτελεσματικό αποτελεσματικός. Και γι' αυτό η διαφάνεια είναι σημαντική, διότι θα μεταθέσει από μια πολύ σε υψηλό βαθμό συγκεντρωμένη αγορά ε, μεγαλύτερη προσπερασιμότητα για άλλους συναλλασσόμενους. Πολλοί μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σήμερα σε τέτοιες αγορές. Ανησυχώ λοιπόν για την επικέντρωση και συμπίκνωση τέτοιων ε, δραστηριοτήτων σε λίγα ιδρύματα ή σε λίγου εμπλεκόμενου. Η τελευταία ανησυχία είναι το clearing houses, τα συμψηφιστικά όργανα. Τώρα, σήμερα, εξαρτώνται αυτά τα όργανα από τους κύριους εμπλεκόμενους που έχουν και πριτανεύοντα ρόλο, δεσπόζοντα ρόλο γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ήθελα να αποφύγω καθόλου την ερώτησή σας ε, σκεπτόμαστε και προσεγγίζουμε σε μεγάλο βαθμό με τον ίδιο τρόπο αυτά τα θέματα πιστεύω. Ερώτηση για τον πρόεδρο Ομπάμα και την λέσχη των 20. Εγώ περισσότερο βρίσκομαι εδώ για να αναφέρω για τα θέματα παραγόγων ε, σε σχέση με αυτές τις δράσεις όσον αφορά την συνάντηση της λέσχης των 20 και όχι μόνο σε σχέση με το τι σκέπτεται κάποιος από την κυβέρνησή μας αλλά και το, τους ε, βουλευτές μας. Πώς μπορούν αυτού του είδους ε, οι πλατφόρμες ε, να ρυθμιστούν. Πώς να υπάρχει κεντρική ρύθμιση από πλευρά συμψηφιστικών αρχών υπήρχε κάποια κίνηση σε σχέση με κάποιους να γίνουν κάποιες ε, ε, ε, ας το συνοδευτικές δράσεις. Δεν θέλω καθόλου να αποφύγω την ερώτηση για τα hedge funds και, και τα παράγωγα. Η δική μου αρμοδιότητα είναι αυτή για τη ρύθμιση αυτών των αγορών παραγωγών Σημερίζεστε την άποψη θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει συμψηφιστικό όργανο και στην Ευρώπη. Ο μιλητής, ναι, σε αυτό υπό τους όρους των συμψηφιστικών αρχών Νομίζω είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί αλλά και οι Ασιάτες ρυθμιστές θα έχουν αυτές τις πληροφορίες από πλευράς ε, συμψηφιστικών οργάνων όπου και αν βρίσκονται. Αν καταλήξουμε με γεωγραφικούς προσδιορισμούς έναν τέτοιο συμψηφιστικό φορέα στην Ευρώπη, έναν αλλού, θα πρέπει παρόλα αυτά πάλι ε, και ένα στην Ασία, θα πρέπει εμείς στη ΣΥΠΑ να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Αν έχουμε την ε, εντολή αυτή, παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουμε σημεριζόμενο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και διατάξεων. Γιατί αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να δρουν σε άλλη νομοθετική περιφέρεια. Θα ε, ε, ξετυλίγουν τις αρμοδιότητες τους αλλού. Το να έχουμε μια ρυθμιστική αρχή στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι καλύπτει το πρόβλημα επαρκώς. Πρέπει να είμαστε διασυνδεδεμένοι σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Δεν ρυθμίζουμε όσον αφορά το Trade Depository που ήταν στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων και δράσεων δεν ε, έχει ρητά τέτοια αρμοδιότητα. Δεν υπάρχουν ε, νομοθετικές προτάσεις σε σχέση με αυτή τη δράση. Υπάρχουν όσον αφορά τη ρύθμιση ε, συμψηφιστικών οργάνων. Δεν έχουμε όμως το, συμψηφιστικό κύριο όργανο το οποίο χρειάζεται. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό. Ευχαριστώ. Um, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πασκάλ μετά η Κατρίν παρακαλώ. Yes. Να επανέλθω στην πρότασή σας σχετικά με τον περιορισμό των θέσεων σε ό,τι φορά τα παράγωγα. Νομίζω ότι αυτό εφαρμόζεται σε κάποιες ε, αγορές στις ΗΠΑ. Θα μπορούσατε να πείτε κάτι παραπάνω σχετικά με το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο παρόμοιο σύστημα και τι είδους αρχή θα είναι αυτή που θα λαμβάνει τις αποφάσεις θα θα εφαρμόζεται μόνο στι ΗΠΑ ε, διασυνοριακά πώς. Και η Κάθριν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο εξετάζεται το ζήτημα. Είπατε ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι σχετικά με το εάν υπήρξε μια αλλαγή κουλτούρα στην ε, Wall Street ε, μετά από τα γεγονότα και σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, λογιστικής ε, θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια συμφωνία χωρικά και με το θέμα της ευθύνης και το ποιος είναι υπόλογος για τη λογοδοσία. Ναι, έχουμε κάποιες αρχές για θέματα που η Γεωργία είναι η SFTC που έθεσε κάποια όρια, κάποιου περιορισμού σχετικά με την κατοχή αυτών των ε, παραγόγων για προϊόντα γεωργικά ή για άλλα είδη πρώτης ανάγκης. και φυσικά προσπαθήσαμε να πετύχουμε να υπάρχει μια ποικιλία ε, συναλλασσομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα credit defaults και τα swaps, καταδίσαμε κάποιους κανόνες και τα credit for swaps, τα CDS, τα Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης, εξετάζοντάς τα, παρατηρούμε ότι ε, μπόρεσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τώρα πώς το πετύχαμε. Δώσαμε τις αρμοδιότητες στην κατάλληλη αρχή. Τώρα για το αν έβαλε μυαλό η Wall Street, ε, τι να σας πω. Ελπίζω. 18 χρόνια εμπειρία είχα στην Wall Street. Αλλά ξέρετε ότι είναι δύσκολο να μην διαπράξει κάποια σφάρματα ο άνθρωπος έχουν ε, και κάποιες υποχρεώσεις όλοι ε, αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στους μετόχους, τη ε, μεγιστοποίηση του κέρδους κλπ. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου, να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε φυσικά είναι να προστατεύσουμε τους φορολογούμενους, ειδικά τώρα από την θέση την οποία κατέχουν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποια σύγχυση στα πράγματα. Νομίζω πως συνεχίζει να υφίσταται κίνδυνο στο όλο σύστημα. Εγώ συνεργάστηκα με την Μέρη Σαπύρο στενά τον ε, τελευταίο καιρό. Δεν θα πρέπει να την ε, επικρίνουμε. Καταβάλει κάθε προσπάθεια και άλλα όργανα συνεργάζονται με την ε, Μέρη Σαπύρο και η FCC ότι ο στόχος μας είναι κοινό, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις. Η κυρία Άννη Ποδηματά και μετά η Βίκη παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για τις απαντήσεις σας. Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση στις Ηνωμένε Πολιτείες για ενδεχόμενη δημιουργία αρχής προστασίας καταναλωτών. Δεν ξέρω αν δεν πρόλαβα κάτι γιατί καθυστέρησα να έρθω, αλλά για μας είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και θα μπορούσε να περάσει το μήνυμα στους φορολογούμενους ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα συμφέροντά τους και ότι τα συμφέροντα του καταναλωτή είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις μεταρρυθμίσεις και για καλύτερη ρύθμιση των αγορών. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιδέα αυτή. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Και βεβαίως, επειδή γνωρίζουμε ότι υπήρξαν και πολλές αρνητικές αντιδράσεις για την ιδέα αυτή, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ακόμη ελπίδες ότι θα καταλήξουμε σε μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτών. Δεύτερη ερώτηση. Αναφέρατε ότι τα παράγωγα έπαιξαν κάποιο ρόλο στην οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και υπάρχει και κάποια συζήτηση συγκεκριμένα για την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να υποθούν εδώ. Η Ελλάδα, αλλά όχι μόνο η Ελλάδα, γιατί υπήρξε μια κοινή επιστολή από τους ε, κυρίους και κυρίες Μέρκελ, Σαρκοζή, Γιούνκερ και τον Έλληνα Πρωθυπουργό του κύριο Παπανδρέου που ζήτησαν σαφείς κανόνες για τα CDS και απόλυτη απαγόρευση των CDS όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Πιστεύετε ότι αυτά τα γυμνά CDS είναι μία θεμητή επιλογή όταν μιλάμε για το δημόσιο χρέος. Ευχαριστώ, Δίκη. Ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας σήμερα εδώ γιατί πολλοί έχουν πει ότι πρέπει να κοιτάμε την παγκόσμια αγορά και να έχουμε παγκόσμιο συντονισμό οπότε είναι χρήσιμο να ακούμε την άποψη πέραν του Ατλαντικού. Υπήρξε μία έρευνα αυτή τη βδομάδα που έδειξε ότι τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά κέντρα είναι από κοινού Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Κάτι που απογοήτευσε λίγο το Λονδίνο, εν πάση περιπτώσει. Όμως, εσείς τι κάνετε προκειμένου να συνομιλήσετε με όσους βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αν θέλουμε κάτι παγκόσμιο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και αυτό. Επίσης νομίζω ότι η αναλογία που κάνατε μεταξύ CDS και ασφαλιστικών προϊόντων είναι πολύ χρήσιμη. Και βεβαίως, όπως ακριβώς και με τις ασφάλειες, γνωρίζουμε ότι έχουμε τους αγοραστές και τους πολιτές του κινδύνου και πρέπει να δούμε τη διαφορετική θέση του καθενός. Αν για παράδειγμα εγώ αυτή τη στιγμή είχα συναλλαγές με με ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να με ενδιέφερε να αγοράσω ασφάλεια γενικά για την Ελλάδα. Όμως κάτι τέτοιο μπορεί να ήταν διαφορετικό αν το βλέπαμε από την πλευρά του πολιτή του κινδύνου. Τώρα, ακούω από πολλούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ε, στη δικιά μας πλευρά του Ατλαντικού για το πώς μπορούμε να βρούμε λύση και τους ακούω να ζητούν εξαιρέσεις όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για τους βασικούς πελάτες τους. Άρα πολλές ε, προσπάθειες lobbying όσον αφορά τις εξαιρέσει αφορούν τις ε, μεγάλες εταιρείες. Και αυτοί θέλουν να μειώσουν το κίνδυνό τους. Τώρα, όντως ε, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με τον αριθμό των οργανισμών συμψηφισμού, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία κατακαιρματισμένη αγορά και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο σε επίπεδο διεπαφής παρόλο που θα μείωνε τους κινδύνους υπερβολικής συγκέντρωσης. Είναι λοιπόν κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Επίσης, μιλήσατε για τα χρηματιστήρια διαφάνεια, καλύτερη τιμολόγηση, μείωση του κινδύνου. Εμείς έχουμε ασχοληθεί πολύ με το πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των χρηματιστηρίων προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και να βελτιωθεί η τιμολόγηση. Βεβαίως το θέμα είναι δύσκολο και δεν μπορούμε απλά να πούμε ότι ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε καλύτερες τιμές. Και αν και βεβαίως δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μονοπόλια. Ευχαριστώ. Υπενθυμίστε μου αν ξεχάσω κάποια ερώτηση. Όσον αφορά την αρχή προστασίας καταναλωτών, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τη ΣΥΠΑ και συμμερίζεται την άποψή μου η κυβέρνηση ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές γιατί ήταν τμήμα της κρίσης τα παράγωγα αλλά ένα τμήμα της κρίσης ήταν και τα στεγαστικά δάνεια, οι υποθήκες. η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε την ε, πρόταση της κυβέρνησης για την αρχή προστασίας των καταναλωτών. Τώρα, στο πακέτο που περνάει από τη Γερουσία ακόμη συζητάτε το θέμα. Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ανεξαρτησία. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές από τις ε, προστατευτικές δικλίδες βρίσκονταν εντός ε, των ε, ρυθμιστικών αρχών των χρηματραπεζών και πολύ συχνά το πρόβλημα ήταν ότι μας ενδιέφεραν πρώτα οι τράπεζες και μετά οι πελάτες των τραπεζών. Εγώ προσωπικά εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Όμως έχει συζητηθεί πολύ, ειδικά από τις εμπορικές τράπεζες, όχι τόσο από όσους ασχολούνται με τα παράγοντα. Όσον αφορά τα CDS, υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σαφής μεταρρύθμιση για τα CDS όπως και για όλα τα παράγωγα. Διάβασα την επιστολή που αναφέρατε. Είναι σημαντικό να υπάρχει τη δυνατότητα η ρυθμιστική αρχή να αποφεύγει τη χειραγώγηση και να θέτει όρια. Τώρα, όσον αφορά μια πιθανή κατάργηση των γυμνών CDS, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το κάνει κανείς αυτό. Αλλά ακόμη και αν μπορούσαμε να το κάνουμε, εγώ πιστεύω ότι η κερδοσκόπη είναι κομμάτι της αγοράς. Και είναι πολύ δύσκολο να διαπιστώσουμε αν κάποιος κάνει απλά hedging, κάλυψη του κινδύνου ή αν κερδοσκοπεί. Άρα χρειαζόμαστε κανόνες κατά της χειραγώγησης της αγοράς. Χρειαζόμαστε και περιορισμούς για τις θέσεις. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά από μια διαφανή διαδικασία συναλλαγής ε, των CDS. Χαίρομαι που αναφέρατε και το MIFID ξανά. Αυτά τα παράγωγα θα μπορούσαν να έρθουν σε κεντρικές ε, πλατφόρμες και θα μπορούσαν να, να λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς για το υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς. Νομίζω ότι για τα CDS γενικά έχουμε να κάνουμε με τυποποιημένες τιμές, είτε αφορούν χώρα για δημόσιο χρέος, είτε οτιδήποτε άλλο. Όσον αφορά τον παγκόσμιο συντονισμό, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε πολλά. Είχαμε περίπου 20 χώρες που συζήτησαν, η Ιαπωνία, Ινδία, Μεξικό και ορισμένες ρυθμιστικές ε, ρυθμιστικοί οργανισμοί. Όλοι μας μαζί, αν και δεν είχαμε την Κίνα. Το σίγουρο είναι ότι όλος ο κόσμος προσβλέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα γίνει κάπου αλλού. Έχουμε λοιπόν επιρροή στις τρίτες χώρες, έστω με κάποιες εξαιρέσεις. Όσον αφορά τώρα τους οργανισμούς συμψηφισμού, δεν θα έπρεπε να υπάρξουν περιορισμού για τις ε, γεωγραφικές θέσεις. Υπάρχει μια πρόταση για το Λονδίνο. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καλό διάλογο με αυτούς. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα έχουμε καλή ρύθμιση και από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες, γιατί εμείς θεωρούμε ότι εμείς ως Αμερική θα πρέπει να μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες αυτού του οργανισμού, όπου και να βρίσκεται, αν λοιπόν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε νομίζω ότι οι συγκεκριμένες γεωγραφικές εντολές θα αυξήσουν και όχι θα μειώσουν το κίνδυνο. Αυτά και ελπίζω να μην ξέχασα κάποια ερώτηση. Βίκη, για το σημείο αυτό συμφωνείτε ότι τα ασφαλιστικά μπορούν να έχουν ένα διαφορετικό προφίλ κινδύνου όσον αφορά σε σχέση με το CDS. Νομίζω ως αναλογία αυτό απάντηση. Νομίζω ότι σε σχέση με τα ασφαλιστικά. Πρέπει να υπάρχει σαφής αρχή από τους ρυθμιστές για κεφαλαιακές ανάγκες ε, όσον αφορά τέτοιες συναλλαγές και τις τράπεζες που πολλούν ε, CDS. Είναι διαφορετικό το θέμα από, σε, σχέση με τα επιτόκια. Μπορεί κανείς ε, με υπολογισμό αναλογιστικό να το δει. Είναι όμως ένας ασυνεχής κίνδυνος αυτός, ένας εκπεριτροπής εμφανιζόμενος κίνδυνος. Από πλευρά των αγοραστών όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε οι κεφαλαιακές αυτές προδιαγραφές σε σχέση με τις τράπεζες που αγοράζουν CDS όσον αφορά και την, ε, ε, τις κεφαλαιακές ανάγκες, το capital arbitrage. Το η AIG τι έκανε, έδινε το όνομά της ε, σε πολλές τέτοιες συναλλαγές και είχαν και μείωση των δαπανών οι τράπεζες στην Ευρώπη αγοράζοντας CDS. Από αυτό μπορεί να αγοράσει κανείς, να, να συναγάγει κανείς συμπεράσματα όσον αφορά την διαχείριση κεφαλαίων όσον αφορά την, τον δανεισμό ενός ονόματος από μια τράπεζα για να γίνουν τέτοιες συναλλαγές από άλλους. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τις ακόλουθες παρεμβάσεις και θα ακολουθήσει και ο Σβέν. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμμερίζομαι το γεγονός ότι η διαφάνεια είναι ένα θέμα θεμελιώδους σημασίας και γι' αυτό είναι απαραίτητο βήμα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Η διαφορά σε σχέση με την κερδοσκοπία όμως είναι ότι σε σχέση με τις συναλλαγές των κερδοσκόπων, στις συναλλαγές δεν συμμερίζονται, δεν συμμετέχουν μόνο κερδοσκόποι, αλλά έχουμε και συναλλασσόμενους της πραγματικής, οικονομία οικονομίας. Και σε σχέση με όσους εμπλέκονται σε αυτό το πλαίσιο, με την κερδοσκοπία υπάρχει στρέβλωση και μεγάλη, θα έλεγα, ε, αλλαγή πραγμάτων, ευμετάβλητο ε, χαρακτήρα όταν έχουμε τους συναλλασσόμενους όμως που δεν έχουν την διακάλυψη. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα που είναι σημαντικά σημαντικές για την πραγματική οικονομία το πρώτο. Τι γίνεται. Να αποφύγουμε δεύτερον αυτή τη δυσαναλογία μεταξύ των κινδύνων που επομίζονται οι συναλλασσόμενοι όσον αφορά ε, τέτοιες δράσεις ε, στην ε, πραγματική οικονομία. Το να περιοριστούν αυτά τα πλαίσια είναι σημαντικό αλλά δεν επαρκεί πρέπει να υπάρξει σημαντική διασύνδεση μεταξύ αγορών, μεταξύ των παραγόγων για παράδειγμα και των πραγματικών συναλλαγών, μεταξύ των εγγυήσεων που θα ε, ε, καλύπτουν τις κανονικές συναλλαγές θα πρέπει να θεσμιστούν, θεσμοθετηθούν συγκεκριμένες ε, προδιαγραφές για την κάλυψη αυτών των συναλλαγών. Και αν έχουμε ένα φόρο για τις συναλλαγές, ένας τέτοιος φόρος στις οικονομικές, τέτοιες χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα μπορούσε να συνεισφέρει στον να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των αγορών. Ευχαριστώ. Uh, Εγώ από πλευρά μου έχω κάποιε σύντομε ερωτήσει. Πρώτον, με εξέπληξε κάπω το ότι είπατε ότι θα ήταν δύσκολο, λέει, να απαγορευτούν κάποια προϊόντα. Από την άλλη όμως πλευρά, είσαστε, λέει, πολύ πιο αισιόδοξο να περιοριστούν ε, οι όγκοι συναλλαγών, size of positions μου δημιουργεί κάποια σύγχυση το ότι είσαστε περισσότερο αισιόδοξο για το ένα, λιγότερο αισιόδοξο για το άλλο. Μπορείτε κάπω να επεξηγήσετε την ε, τοποθέτησή σα σε αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Και σα ζητώ να είσαστε το δυνατόν ομότερο ε, και κατηγορηματικό. Υπάρχουν τομεί όπου η δράση ρυθμιστικών ή εποπτικών ε, τέτοιων αρχών στην Ευρώπη ή σε κάποια κράτη-μέλη στην Ευρώπη δίνουν ε, ε, καθιστούν τη δουλειά σας στη ΣΥΠΑ δυσχερέστερη. Τι γίνεται σε σχέση με σας ε, στη ΣΥΠΑ λόγω αυτών, λόγω ανταγωνισμού για παράδειγμα από την Ευρώπη, ότι είναι πιο δύσκολο για σας να καταλήξετε με νέες ρυθμιστικές διατάξεις ή αυστηρότερη εποπτεία στην πραγματική εφαρμογή των κανονισμών. Τρίτον, αν δούμε την παγκοσμιοποιημένη κατάσταση σήμερα, υπό το δικό σας πρίσμα, Ποια μέσα έχει, έχουν οι ΙΠΑ ή έχουν οι Ευρωπαίοι ώστε να καταστήσουν πιο θελκτικές, πιο ελκυστικές, ε, για να το πω αυτό ήπια, για τρίτες χώρες το να αυξήσουν και εκείνες τις εποπτικές και ρυθμιστικές τους ε, δραστηριότητες. Επειδή πολλής λόγος γίνεται βλέπετε για την ανάγκη παγκοσμιοποιημένου εναρμονισμού ή ε, συνεργασίας, παγκόσμιας συνεργασίας. Από την άλλη όμως πλευρά, αν αυτά είναι ολολόγια μόνο, αυτό μπορεί να οδηγήσει στον χαμηλότερο δυνατό παρονομαστή ως επίπεδο για την εποπτεία και ρύθμιση. Ερώτηση λοιπόν να ληφθούν από χωρίς ε, να υπάρξει αυστηρός προστατευτισμός βέβαια, χωρίς να καταλήξουμε σε προστατευτισμό, αλλά οδηγώντας σε ισχυρά κίνητρα για τρίτες χώρες να αυξήσουν τις ρυθμιστικές τους προσπάθειες και τις δικές τους εποπτικές προσπάθειες. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Um, Αντίστροφα θα απαντήσω με την τελευταία ερώτηση πρώτα που ε, αντυχεί στα αυτιά μου ακόμα. Υπάρχει πάντα μια πρόκληση όταν συνέρχονται η και η Ευρώπη, άλλε χώρες και άλλε ε, νομοθεσίες και ρυθμιστικές αρχές να κάνουν κάτι. Όμως η κύριη μοχλή μέσα που έχουμε στα χέρια μας είναι εφόσον πρόκειται για παγκοσμιοποιημένε αγορές ε, που, ε, και συναλλαγές που ρυθμίζονται είτε από πλευράς ευρωπαϊκών αρχών είτε τον είπα να πει κανείς σε μια μεγάλη τέτοια χρηματοοικονομική τράπεζα ότι σας ε, προσεγγίζουμε από την Consolidated Group ή να δούμε εδώ την ε, εξατομικευμένη ε, νομική ας το πω έτσι εγκύτητα και το τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος και να πει ε, εφόσον συμβαίνει αυτό εδώ και με παρακολουθούν εκ του σύνεγγις θα μεταφερθώ αλλού. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το αποκαλέσει regulatory arbitrage. Αλλά αν όμως οι ρυθμίσεις αφορούν μια ολόκληρη ομαδοποιημένη, μια ολόκληρη ομάδα άσχετα από το που έχει την έδρα της ε, και για τους 14 ε, μεγαλύτερους που αναφερθήκαμε πιο πριν. Ο άλλος μοχλός που έχει κανείς είναι πρόσβαση στους επενδυτές, ε, access to investors ώστε τελικά στην αγορά αγαθών για παράδειγμα όσον αφορά τα αγαθά τα προϊόντα γεωργίας π.χ. Αν όμως θέλει κανείς να προσφέρει trading screen έναν έλεγχο από πλευράς είπα και να έχουμε ένα τέτοια, μια τέτοια ε, ας το πω έτσι εξέταση του τι γίνεται από πλευράς αυτών των συναλλαγών π.χ. στο Κάνσας δεν είναι πλήρης αυτή από πλευρά μας αλλά πολύ Δουλειά πρέπει να γίνει και από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρώπη. Ρωτήσατε για κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν. Έχουμε μέλη της Βουλής μας που λένε ότι αν γίνει αυτό στις ε, ΗΠΑ και ε, εμείς περιορίσουμε τη δραστηριότητα αυτών των εταιριών θα πάνε όλοι στην Ευρώπη ή αλλού ενθαρρύνομαι με την αντιμετώπιση την ε, ε, σφαιρική και λέω σε αυτό πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε όλοι τα προβλήματα. Αλλά υπάρχουν ρογμές, ε, χαραμάδες για τους συναλλασσόμενους στο σύστημα που μπορούν να διαφύγουν από εκεί ίσως και να πάνε αλλού και να δράσουν αλλού. Όμως είναι πρόκληση του να δει κανείς το τι έγινε με το CDS. Πρόκληση επίσης του τραπεζικού απόρριτου που αντιμετωπίζουμε σε πολλές τέτοιες συναλλαγές. Πρόσβαση σε πληροφορίες για ρυθμιστικές αρχές για παράδειγμα και περιορισμοί. Θα έλεγα όμως ε, γενικά ότι ο συντονισμός ε, στις προσπάθειες αυτές μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης είναι πολύ θετικός και καλός. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις ε, είναι να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι είναι το hedging έναντι των, της κερδοσκοπίας, speculation πότε κάτι μπορεί να θεωρηθεί γυμνό ή ο ξεκάθαρο CDS, άμεσο CDS. Και τι γίνεται σε σχέση με τα, ακριβώς αυτά τα credit default swaps, τα CDS, έχουμε και position limits, ε, όρια ε, συνολικά συναλλαγών, που δεν είναι το τέλειο εργαλείο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε η ρυθμιστική αρχή να μπορεί να δράσει καλύτερα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μία άλλη κέρια ερώτηση. Τι γίνεται σε σχέση με τη διαφάνεια, που ενώ είναι σημαντική και βοηθά, υπάρχει, δεν σας αναφέρω στο παράθεμα σωστά, αλλά υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τη σχέση των κερδοσκόπων όσον αφορά τις συναλλαγές και τις αγορές. Έχετε δίκιο, υπάρχει πολλής κίνδυνος που εξωτερικεύεται, εξωτερικοποιείται. Η Wall Street και η AIG εξωτερήκευσαν αυτόν τον κίνδυνο όσον αφορά τους πολίτες, τους φορολογούμενους και έτσι ήταν, ας το πω έτσι, ε, ρίχνανε το νόμισμα, κορώνα γράμματα και τα σπασμένα τα πλήρωναν πάντα οι φορολογούμενοι, οι πολίτες. Εδώ θα πρέπει να παρέμβουμε και να υπάρχουν οι ρυθμιστικές αρχές συμψηφισμού, να δράσουν τα clearing houses, ώστε σε περίπτωση τέτοιων ε, ε, συναλλαγών να μπορούν έγκαιρα να παρέμβουν. Δεν είναι όμως δωρεάν όλα αυτά. Δεν μπορεί κάποιος να πει «Α, δεν μπορώ εγώ να δεχθώ υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες». Γι' αυτό έχουμε την πολιτική διαδικασία να επιλέξουν οι νομοθέτες να επιλέξουν τις, ε, να αντιμετωπίσουν σωστά τις δύσκολες προκλήσεις νομοθετικά και να θεσπίσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Και να δούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με τις άλλες συναλλαγές, όπως αφορά τα γεωργικά προϊόντα, έχουμε την Anti-Manipulation Authority, ώστε να ε, μπορέσουμε να αποφύγουμε κερδοσκοπίες όσον αφορά, ε, για παράδειγμα, σιτηρά, κρυθάρι, σιτάρι κτλ. Αλλά παρόμοια προσπαθούμε και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές να μπορέσουμε να δράσουμε δράσουμε παρεμβατικά. Νομίζω απάντησα υπαρκώ. Ευχαριστώ. Όχι, συγγνώμη. Θα έπρεπε να μεταφράσω α, τα όσα είπα σε πιο απλή γλώσσα corner squeeze είναι όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, όταν κάποιος μπορεί να έχει πληθώρα ενός προϊόντος που βρίσκεται υπό περιορισμένη διάθεση, σε περιορισμένη διάθεση, ώστε να μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή από πλευρά σου στις τιμές και στην πώληση. Και αυτό γίνεται βάσει ενός συμβατικού συμβολέου για τη διάθεση αυτών των προϊόντων. Οι Hunt Brothers προσπάθησαν την αγορά, για παράδειγμα, αργύρου να την ελέγξουν έτσι με αυτόν τον τρόπο, αγοράζοντας με επιθετικό τρόπο συμβόλαια futures μελλοντικής ε, ε, ε, εκφοράς για το προϊόν αυτό, για τον Άργυρο. Και βλέπουμε ότι κάτι παρόμοιο είχαμε και στις αγορές φυσικού αερίου πρόσφατα και είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Στην αντίστοιχη περίπτωση είχαμε τέτοιου είδους περιπτώσεις που δίνουν ιστορικά μεγάλης σπουδαιότητας τέτοιες ε, ε, συγκεκριμένες δράσεις. Όταν βλέπουμε ότι squeezer είναι ε, σε περίπτωση σπανίδας ενός αγαθού η διάθεση από πλευρά συναλλασσομένων κερδοσκοπικά. Ευχαριστώ. Επεκτηνόμενο σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν για την απαγόρευση προϊόντων, θα ήθελα να επεκτείνω λίγο πέρα από το CDS, το Credit Default Swap όταν αρχίζουμε να λέμε να απαγορευτούν κάποια προϊόντα ή πρακτικές, είναι δίπλευρη, διμερής η εικόνα. Αφενός υπάρχουν εκείνοι και ίσως αναφερθήκατε σε αυτούς πιο πριν ότι τα εμπόδια, τα προσκόμματα πρέπει να είναι υψηλότερα. Ε, ε, το να επιτρέπει κανείς είναι ευκολότερο όταν δυσκολεύονται λόγω προσκομμάτων ή προδιαγραφών οι συναλλαγές. Κανείς όμως ε, δεν θέλει να κινδυνεύει από τοξικά προϊόντα. Απαγορεύτηκε ο αμίαντος στις οικοδομές ε, και ε, έχουμε όμως τοξικά προϊόντα στα χρηματοοικονομικά. Γιατί να μην απαγορευτούν. Τώρα για την παρατήρησή σας για το CDS είναι τεχνικού χαρακτήρα αυτή η διαφοροποίηση. Η χρήση που γίνεται δηλαδή αυτών των μέσων αυτό που είπατε ισχύει για οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν. Για παράδειγμα για τις συναλλαγές στη Wall Street, στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Ε, όχι υπό την σημερινή σας αποκλειστικά αρμοδιότητα. Έχοντας πείρα 18 ετή στο χρηματιστήριο στη Wall Street, είδατε κάποιες πρακτικές ή μέσα ή προϊόντα που θα έπρεπε να απαγορευθούν. Πρακτικές ή προϊόντα διότι αποσταθεροποιούν και οδηγούν σε στρεβλώσεις. Ευχαριστώ. Uh, Εντάξει, να σας απαντήσω. Είδα πολλά να γίνονται στο, στη Wall Street, στο χρηματιστήριό μας αυτά τα 18 χρόνια. Ακόμα και όταν επαγγελματίες ε, ε, ακολουθούσαν τέτοιες πρακτικές ε, με καλές προθέσεις και νόμιμα, καλ, πολλές φορές διερωτώσουν γιατί να το κάνει αυτός ή ο άλλος αυτό ή το άλλο. Ακόμα και όταν μπορεί ένα δάνειο σε ένα παράγωγο να εντάσσεται, δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό, αλλά γίνονται όλα αυτά επίσης και πάλι. Όσον αφορά το CDS, Credit Default Swaps πάλι, σε σχέση με αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσαμε να ε, προσπαθήσουμε να απαγορεύσουμε τέτοιου είδους πρακτικές. Χειροπιαστά όμως πρακτικά θα, θα έβρισκαν άλλους τρόπους αυτού του είδους ε, τις πρακτικές να τις εκφράσουν και στις, ε, στα ασφαλιστικά συμβόλαια ή αλλού ή αυτές τις πρακτικές. Ή με την αγορά για παράδειγμα συμβολέων, ασφαλιστικών συμβολέων για την αυτιλία, πλοίων, ποντοπόρων πλοίων. Από πλευρά Ευρωβουλευτού η παρέμβαση αυτή αληθεύει. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Υιοθετήσαμε όμω μια διαφορετική προσέγγιση στη ΣΥΠΑ. Μια προσέγγιση που την υποστηρίζω. Οι κερδοσκόποι και οι κερδοσκόποι, αυτό speculators δεν είναι ε, βρυσιά στην, <laughs> στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω πώς το μεταφράζετε στις γλώσσες σας. Ο hedger είναι κάποιος που έχει, ας το πω έτσι, ένα χειροπιαστό αγαθό. Ανάγκη να καλυφθούν κίνδυνοι σε σχέση με αυτό το αγαθό. Πολώντας, για παράδειγμα, ε, σε μια χώρα ή μια χώρα ένα τέτοιο προϊόν. Τους βρίσκει κανείς σε μια αγορά από την άλλη πλευρά και τους αποκαλούμε κερδοσκόπους ή επενδυτές κιόλας. Εκείνο το οποίο είναι αρνητικό είναι όταν χειραγωγούν τις αγορές, όταν κάνουν, ας το πω έτσι, τέτοιου είδους ε, συναλλαγές που στρεβλώνουν τις αγορές. Αυτό είναι αυτό το οποίο συζητείται στην ε, Ευρώπη, η στρέβλωση των αγορών. Δηλαδή, γιατί διαφορετικά αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο θα πήγαιναν αλλού. Λοιπόν, αν πραγματικά επικεντρωνόμαστε σε αυτό, είναι η ίδια πολιτική και από πλευρά τη ΕΥΠΑ, Πώ θα μπορέσουμε να προαγάγουμε ανοιχτέ, διαφανεί, ε, χωρί τρευλώσει και καταχρήσει αγορέ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Διαφοροποίηση δηλαδή επενδυτών από κερδοσκόπους. Αυτό είναι ενδιαφέρον και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Απλά και μόνο θα σας ευχαριστούσα αν κάνατε κάποιο σχόλιο για κάποιο το οποίο έθεσα εγώ ως παρατήρηση πιο πριν. Βλέποντας ότι υπάρχει υπετροφία σε κάποιες ε, χρηματοοικονομικές αγορές. Η ερώτηση για τον φόρο αυτό των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αν θα μπορούσε αυτό να εξεταστεί ως ένα από τα θέματα που θα μπορούσαν να εξεταστούν από τη μία ή άλλη όχθη του Ατλαντικού ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι δεν ομιλώ εξ ονόματος της κυβέρνησης Ομπάμα όταν ε, τίθενται τέτοια ερωτήματα και ζητείτε να απαντήσω επ' αυτών. Έχουμε όμως ε, ε, διάφορα τέλη για τις συναλλαγές στις ΗΠΑ που πληρώνουν την δράση των ρυθμιστικών αρχών. Τώρα, αν το αποκαλείστε φόρο ή όχι, είναι όμως τέλη έχουν, ε, υπάρχει σύσταση να ε, εισπράττονται και σε όλες ε, τις συναλλαγές. είναι ένα μέρος του συστήματός μας. Όλοι πληρώνουμε τις ρυθμιστικές αρχές στη δράση τους με τέτοιου είδους τέλη, οι εισφορές. Δεν νομίζω δεν χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν τις αγορές, έτσι. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα τέλη για να πληρώνεται η, ρύθμ, η δράση των ρυθμιστικών αρχών. Και γι' αυτό γίνεται αυτού του είδους η χρήση. Πρέπει να τεθούν υψηλά αυτά τα τέλη, αν θέλετε να περιορίσετε κάποια δράση. Έχουμε λοιπόν το θέμα του κόστους και της προσέγγισης όσον αφορά τα τέλη που θα έπρεπε για τα securities να ληφθούν υπόψη. Υπάρχει κανείς που δεν καλύφθηκε. Πασκάλ, μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ. Σε σχέση με την προηγούμενη ερώτησή μου για το ζήτημα των περιορισμένων, περιορισμένων θέσεων, αν θέλετε, έχετε κάποια στοιχεία κατά νου και τι εργαλεία διαθέτετε ή προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε. Όχι, δεν έχουμε κατά νου κάποια στοιχεία. Τώρα προσπαθούμε να εξετάσουμε το θέμα. Έχουμε, δώσει κάποιες, ε, έχουμε κάνει κάποιες αναθέσεις, κάποιες εξουσιοδοτήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να συστήσουμε την Επιτροπή τώρα σε ό,τι φορά τα γεωργικά προϊόντα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συναλλασσομένων και με πληροφόρησαν ότι φροντίζουν να μην υπάρχει κανείς που να ξεπερνάει το 10% του συνόλου κλπ. Αν πρέπει ότι αν υπάρχουν, υπάρχει το όριο 10% τουλάχιστον θα υπάρχουν 10 εμπορευόμενοι αυτό το αγαθό. Αλλά σε ό,τι αφορά τα CDS θα πρέπει να το ελέγξουμε. Πρόεδρος. Δηλαδή είναι μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία. Ναι, είναι ιδιαίτερα δυναμική διαδικασία, διότι η νομοθετική διαδικασία είναι και αυτή η δυναμική με τη σειρά τη. Και συχνά χρειάζεται να επέλθει κάποια κρίση προτού να ενεργοποιηθεί. Πρόεδρε, νομίζω το εξαντλήσαμε το θέμα. Προσπαθώ να πω και, κάνω και εγώ μια ερώτηση. Και θα είμαι σύντομη. Ζήτημα επικοινωνίας ανάμεσα στους ρυθμιστές ε, και τα επιμέρους κράτη. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένας διάλογος. Όταν ζητάτε προφορίες για τα για τους συμψηφιστικούς ε, οργανισμούς τότε θα μπορείτε να θα, θα πρέπει μάλλον κανεί να έρθει σε επαφή και να διασφαλίσετε πως ε, τα γεγονότα δεν πρόκειται να επανελειφθούν. Εγώ κοιτάξτε αυτή την διασφάλιση δεν μπορώ να σας την δώσω. Έχουμε αλλάξει κάποιους κανονισμούς. Η AIG ε, δεν ρυθμιζόταν ε, σωστά, δεν υπήρχε καλή εποπτεία, αλλά εάν αυτή η μεταρρύθμιση για την οποία μιλάμε περάσει, τότε θα έχουμε γράψει ιστορία και θα δούμε πως ε, θα υπάρξουν κάποια προστατευτικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν την επανάληψη μιας παρόμοιας κρίσης. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε περάσει την ε, μεταρρύθμιση. Α, μιλήσατε για την επικοινωνία. Ε, η επικοινωνία ήταν πολύ αποτελεσματική. Εγώ στην ε, δουλειά αυτή βρίσκομαι 8-9 μήνες. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά εδώ είχαμε πολύ καλές επαφές με τον Μπάφιν, χάρη με τον συμπιστικό οργανισμό της Γερμανίας. Έχουμε υπογράψει κάποια μνημόνια κατανόησης ε, με το Λονδίνο, την FSA. Εμείς, πάση περιπτώσει συνάψαμε με πολύ καλές ε, συμφωνίες και κάποια μνημόνια κατανόησης ε, τα οποία ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Και τέλος, Διερωτώ με αν θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι σχετικά με το συμψηφισμό και τον ε, ρόλο της ε, ρευστότητας. Όπως είπατε θα υπάρξουν ε, κάποιες διμερείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάποιες ε, εξαιρέσεις ε, προκειμένου να μπορούσαν να καλυφθούν κίνδυνοι. Είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξουν ε, τέτοιες ρυθμίσεις προκειμένου να πετύχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αν έχουμε αυτά τα depositories που είναι πολύ περιορισμένα μία κάθε κατηγορία αγαθού παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να βοηθήσει. Εξαιρετικές ερωτήσεις όλες αυτές. Θα έλεγα ένας μεγάλος βαθμός των αγορών μπορεί να καλυφθεί με εκτιμήσεις 3 τετάρτων 75% των συναγών των αγορών που είναι κάτι στάνταρντ για τους συμψηφισμούς. Πρέπει όμως και για την κεφαλική ρευστότητα να ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό είμαι υπέρμαχος να απαιτούμε αυτά τα trading venues να καλύπτονται έτσι. Όταν έχουμε διαφανή διαμόρφωση τιμών τότε λιγότερο εξαρτώνται οι οίκοι συμψηφισμού από τις πληροφορίες αυτές τι γίνεται ε, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ρόλο να διαδραματίσουν για το τι θα συμψηφίζεται ή όχι. Έχουν σαφή, ε, σαφές εξουσίες οι ρυθμιστικές αρχές να διασφαλίζουν ότι οι αρχές συμψηφισμού δεν θα υπομίζονται με κάτι το οποίο δεν θα είναι δική τους αρμοδιότητα, δεν θα υπομίζονται θέματα εκτός των αρμοδιοτήτων τους. Και υπάρχει μια περίοδος ε, για να ρυθμιστεί, να αποφασίσουμε αν είναι κάτι αρμοδιότητα αυτών των οίκων ή όχι. Για την ανθεκτικότητα και το σθένος. Έχουν καλύτερη, ας το πω έτσι, ε, πληκοδότηση τα σώματα συμψηφισμού. Αυτή τη στιγμή αυτά τα 14 μίζωνα ιδρύματα σε σχέση με τα swaps, αυτό το οποίο κάνουν είναι δρούν και ε, ε, σε κάποιους τομείς όσον αφορά και συμψηφιστικές αρμοδιότητες. Έχουν όμως και άλλες αρμοδιότητες. Η καλύτερη εναλλακτική λύση το 75% να ενταχθεί σε αυτού του είδους οίκου συμψηφισμού και να τους διαχειριζόμαστε με συγκεκριμένους στόχους. Δεν έχω υπόψη να έχουν ε, ε, με αυτόν τον τρόπο αποτύχει τέτοιες πρωτοβουλίες. Για depositories είναι κάτι το οποίο έχει ε, κοινά στοιχεία με αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια σαφής ρυθμιστική αρχή που θα ρυθμίζει την εποπτεία. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε ε, κερδοφόρες τέτοιες δράσεις. Μία από τις προκλήσεις όμως είναι αυτό που είπατε εσείς, να διασφαλιστεί ότι θα θα αποφύγουμε την υπερβολική χρέωση τέτοιων συναλλαγών. Η ανοιχτή ε, διακυβέρνηση, διαφανής διακυβέρνηση είναι μια τέτοια δυνατότητα που μας προσφέρεται για να αποφύγουμε στρεβλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαντλήθηκαν ε, οι ερωτήσεις μας και απαντήθηκαν διότι στα δύο λεπτά που απομένουν δεν, νομίζει, δεν νομίζω να έχει υπάρξει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε που θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί για απάντηση σας εξαντλήσαμε και εσάς εξαντλώντας τις δυνατότητες ερωτήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής και να ευχαριστήσω εσάς Πρόεδρε που ήταν δυνατόν να είμαι εδώ παρόν. Αν υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε κάποιες συμβουλές ή συστάσεις να μας το γνωστοποιήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δοθεί συνέχεια σίγουρα σε, αυτό το, σε αυτή την προσφορά. Σας εκτιμούμε ιδιαίτερα για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, πέντε λεπτών, προτού συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.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 Εντάξει, να το αποφασίσουμε. Καθίστε παρακαλώ για να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα μας. Πριν περάσουμε στην επόμενη ακρόαση όμως, θα επανέλθω στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης που την, δεν την έκανα προηγουμένως και πρέπει να γίνει αυτό επισήμως. Να υποθέσω ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη για το υπόλοιπο της συνεδρίασης σήμερα και αύριο. Ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την ακρόαση για την ε, διασυνοριακή διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα. Έχουμε τέσσερις ομιλητές και όπως συνήθως θα κάνουν ο καθένας παρουσιάσεις που θα διαρκέσουν το περισσότερο 10 λεπτά και μετά θα περάσουμε σε ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα... Θα ήθελα να σας συστήσω τους ομιλητές και να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους. Έχουμε τον Στάνισλαβ Κλούζα, πρόεδρο της Πολωνικής ε, Οικονομικής Ελεγκτικής Αρχής, την Κάρμιν Λαμάντα, Senior Executive Vice President και μέλος ε, της Διαχειριστικής Επιτροπής της Unicredit, τον ε, Dirk Schoenmaker, πρίτανη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ντούιζαμπεργκ και την, τον Ριμ Αγιάντη από την Φινιούζ Σέψ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Βλέπω και ένα σημείωμα που με ενημερώνει ότι διανέμονται αυτή τη στιγμή κάποια αρχεία, κάποια χαρτιά που θα έχετε ευτυχώς στη διάθεσή σας. Εγώ τώρα θα αποχωρήσω από την Προεδρία, θα αναλάβει ένας από τους αντιπροέδρους και θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του Στάνισλαβ Κλούζα. Good morning, ladies and gentlemen. I would like uh, ε, ε, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση για τις εμπειρίες της Πολωνικής Ελεγκτικής Αρχής όσον αφορά την διαχείριση της κρίσης, ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχουμε λίγο καιρό στη διάρκεια διάθεσή μας, οπότε θα είμαι σύντομος. Ελπίζοντας ότι θα έχουμε και χρόνο στη συνέχεια για συζήτηση, όπου ίσως μπορέσω να κάνω κάποια περισσότερα σχόλια. Θα ήθελα να μιλήσω καταρχάς για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, τον καταμερισμό των ευθυνών όσον αφορά τις τράπεζες. Δεύτερο θέμα είναι το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη προς τα κράτη-μέλη όσον αφορά την διαχείριση των κρίσεων. Ξεκινάω με την πρώτη διαφάνεια που ίσως προκαλέσει λίγο αλλά δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα βασικό ερώτημα. Ποιος πρέπει να πληρώσει για τις τράπεζες που χρεοκοπούν. Αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό γιατί η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο κάτι που συνέβη στο παρελθόν, είναι κάτι που θα πρέπει να προβλέψουμε και να προδικάσουμε και για το μέλλον. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος θα πληρώσει για την επόμενη κρίση. αυτή τη στιγμή για την κρίση γενικά πλήρωσαν οι φορολογούμενοι. Μπορούμε να γενικεύσουμε περισσότερο ή λιγότερο, όμως σε γενικές γραμμές αυτή τη φορά πλήρωσαν κυρίως οι φορολογούμενοι. Μπορούμε επίσης βεβαίως να πούμε ότι πάντα οι φορολογούμενοι θα είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την κάλυψη οποιασδήποτε κρίσης. Ας δούμε όμως την επόμενη κουκίδα. Ένας νέος ορίζοντας. Ένας δεύτερος υποψήφιος υπεύθυνος. Αν δείτε τις τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπετε επιδείξει, υποδείξεις ότι θα μπορούσε να αφορά γενικά την διαδικασία μεταφοράς των αγαθών από και προς θυγατρικές. Αυτό όμως τελικά θα δημιουργούσε τη δυνατότητα μετατόπισης ευθυνών σε τοπικούς πιστωτές, τοπικά ταμεία εγγυήσεων και ίσως να χρειαστεί να πληρώσουν σε τοπικό επίπεδο κάποιοι για διεθνή προβλήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λύση με βάση τους ε, βασικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πω ότι θεωρώ ότι αυτή η λύση ίσως να αντίκειται σε κάποιες ευρωπαϊκές συμβάσεις και κανόνες. Επίσης, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να μειώσει την ηθική επιληψιμότητα των διαδικασιών αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλήγουμε σε μία τρίτη λύση, ένα τρίτο δρόμο και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να επικεντρωθώ σε αυτή την τρίτη λύση και να εντοπίσω τα βασικά στοιχεία αυτής της λύσης προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τα συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πώς μπορούμε να καλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε την κρίση και πώς θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε συστήματα εγγύησης των καταθέσεων DGS έτσι ώστε και να μπορέσουμε να πληρώσουμε για την κρίση αλλά και αν μπορούμε να προλάβουμε την κρίση μειώνοντας αυτή την ηθική επιληψιμότητα, τον ηθικό κίνδυνο, moral hazard. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σαφή ρύθμιση. Αν δείτε πόσο κόστισε η διάσωση το 2008, βλέπουμε ότι θα ήταν καλό να είχαμε καλές λύσεις που να μειώνουν τον κίνδυνο. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να έχουμε σημαντικό κίνδυνο και τεράστιο κόστος. Εδώ περνάμε στο ρόλο του κράτους. Το κράτος θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το μέγεθος των δραστηριοτήτων και επίσης να μην έχουμε το μοντέλο των ιδιωτικών κερδών, αλλά όταν έχουμε ζημιές, οι ζημιές είναι δημόσιες. Προκύπτει βέβαια εδώ το ερώτημα του ποια κριτήρια θα θέσει το κράτος για το μέγεθος που θα χρειάζεται να έχει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να έχουμε αυτό το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά αυτό της ρευστότητας. Δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ, όμως στην Πολωνία χρησιμοποίησαμε ένα, μια πράξη νομοθετική για ελεκτικά θέματα που αφορά την ρευστότητα, τους κανόνες ρευστότητες. Δεν προέκυψε από κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία, όμως θεωρήσαμε ότι μέσω αυτών των απαιτήσεων για ρευστότητα που είχαμε εφαρμόσει, είχαμε πολύ περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης της κρίσης και επίσης δυνατότητες αποφυγής ή μη τόσο γρήγορης εξάπλωσης της κρίσης. Και βεβαίως η ρευστότητα καθορίζει και τη δυνατότητα Κάλυψη των υποχρεώσεων. Και μας ενδιαφέρει βεβαίως πόσο μεγάλες είναι οι υποχρεώσεις σε σχέση με το κεφάλαιο και πόσο μεγάλη είναι η ρευστότητα σε σχέση με την κάλυψη του κεφαλαίου. Με βάση τους κανόνες μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα των Ιδρυμάτων έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν τουλάχιστον 30 ημέρες εν μέσω οικονομικής κρίσης αν υπάρξει κάποια στιγμή τέτοιου είδου πίεση. Περνάω στο τελευταίο διάγραμμα που αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ε, ευρωπαϊκή συζήτηση όσον αφορά τα συστήματα εγγύησης. Θεωρώ ότι αυτό το διάγραμμα μας επιτρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή σύγκριση. Βλέπετε το μέγεθος των καταθέσεων στις μεγάλες τράπεζες και ποιες από αυτές τις μεγάλες τράπεζες είχαν προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Διαπιστώνουμε ότι ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο αν είχαμε μια πραγματικά παγκόσμια κρίση. Οπότε το θέμα είναι να αποφύγουμε την κρίση, να διαχειρίσουμε την διαδικασία έτσι ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους ε, χειραγώγησης των αγορών. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το πώς θα μπορούσαμε να μοιραστούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις συνέπειες της κρίσης. Ειδικά αν πρόκειται για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν προβλήματα. Αν συνέβαινε μια τέτοια κατανομή ευθυνών θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ηθικής επιληψιμότητας, το moral hazard. Αν χρησιμοποιούσαμε ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων για όλη την Ευρώπη, αυτό θα ήταν κακός σχεδιασμός και θα μπορούσε να αυξήσει εν δυνάμει τους κινδύνους. Γιατί ναι μεν θα προσέφερε κάποια κάλυψη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά θα τους έδινε τη δυνατότητα να εξακολουθούν να κάνουν χειραγώγηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε εσάς κύριε Κλούζα. Τώρα ο κύριος Κάρμιν Λαμάντα θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ που με καλέσατε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην προηγούμενη θητεία μου όταν δούλευα στην Τράπεζα της Ιταλίας όπου διαχειρίστηκα σημαντικές κρίσεις ε, του παρελθόντος. Θα ακολουθήσω το κείμενο των διαφανειών που σας ε, έχω διανύμει. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι σημαντικό. Αυτό το οποίο πρέπει να υλοποιήσουμε ένα σύστημα ευρωπαϊκής εποπτείας ε, πολύ ισχυρό με μια κεντρική αρχή ιδιαίτερα ισχυρή και ένα σύστημα εποπτείας ε, στα κράτη-μέλη υψηλής ποιότητας για να προλαμβάνουμε τις κρίσεις και να τις διαχειριστούμε με το, λιγότερο, με το περισσότερο χαμηλό κόστος. και Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα εποπτείας και να γίνονται συμφωνίες χωρίς να υπάρχουν χαμένοι. Ευχαριστώ αυτό ένα προήμιο τώρα. Γιατί μιλάμε, μιλάμε για ε, τραπεζικούς ομίλους όπως δική μας, ε, στο οποίο ηγείται μια holding και έχει πάρα πολλές ε, τράπεζες σημαντικού μεγέθους στις χώρες μέλη. Αυτό είναι ένα μέσο ιδιαίτερα χρήσιμο για την οικονομική ολοκλήρωση. Είναι ένα μέσο το οποίο πραγματικά υλοποιεί την ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δώσει σταθερότητα και στα διάφορα και με τους διάφορους μηχανισμούς ε, που εφαρμόζουμε. Έχουμε συνάψει συμφωνία με το, Ευρωπαϊ... με το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την οικονομική σταθερότητα. Εάν αυτά είναι θετικά στοιχεία, δεν θα... πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα πρέπει να καταστρέψουμε τα ωφέλη τα οποία έχουμε προκαλέσει. Δηλαδή να κάνουμε να οπισθοδρομήσουμε, να επιστρέψουμε λοιπόν στον προστατευτισμό που θα είναι η καταστροφή του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματο. Η Κομισιόν έκανε σημαντικέ προτάσει για την υλοποίηση αυτή τη εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ πάντω ο δρόμο προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτή την ισχυρή δομή για την πρόληψη και περιορισμό των κρίσεων θα πρέπει να ακολουθήσει τις συζητήσεις οι οποίες ε, εξελίσσονται στο Κοινοβούλιο που είναι πολύ σημαντικές και δαραλές. Τώρα, πότε αντιμετωπίζουμε κρίση, πότε μια τράπεζα βρίσκεται σε κρίση. Βρίσκεται σε κρίση όταν η αγορά τη αφαιρεί την εμπιστοσύνη τη. Δεν είναι πια σε θέση να συλλέξει καταθέσει και να έχει ρευστότητα, δεν μπορεί να διατηρήσει μια υψηλή ρευστότητα, κάτι που είναι απαραίτητο. Κάτω αυτέ τι προποθέσει λοιπόν, που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης ρευστότητα, η τράπεζα ενώπιον αυτή τη κρίση σύμφωνα με πρόσφατη εμπειρία, τι κάνει ε, προσπαθεί να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία για να διατηρήσει την ρευστότητα. Αυτή η πώληση τη ε, περιουσιακών στοιχείων είναι αυτό το οποίο καταστρέφει την τράπεζα, διότι περιορίζει την, ε, την αξία τη και <clears throat> όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει επιρροή και στην περιουσιακά στοιχεία των άλλων τραπεζών. Λοιπόν, ενώπιν μια τέτοια κατάσταση τι θα πρέπει να γίνει άμεσα όταν δεν υπάρχει πλέον αυτή η εμπιστοσύνη και είναι δεδεωμένο, οι αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν ε, θέτοντας στο συμβούλιο, το ειδικό Συμβούλιο της Τράπεζας ε, άτομα τα οποία θα διαχειριστούν την κρίση το να διαχειριστεί κανείς την κρίση εκ των έσω είναι σημαντικό για να ξεφύγουμε από τα προβλήματα που ανέφερε προηγούμενο κ. Κλούς ότι δηλαδή κάποια στοιχεία να μεταφέρονται από μια χώρα σε άλλη και αυτό να επηρεάσει την, την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η, λοιπόν, ένας αποτελεσματικός έλεγχος και αποτελεσματική διαχείριση θα αποφύγει μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ε, μια αρχή η οποία θα είναι ικανή να το πράξει. Λοιπόν, ποιοι είναι η λόγοι, ποια είναι η λογική που θα πρέπει να διέπει την κρίση. Ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε την ε, δημοσιονομική σταθερότητα, να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα και να αποφύγουμε να πληρώσει υψηλό κόστο ο φορολογούμενο. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία μπορούμε να επιλύσουμε και τι ε, διαφορές ε, που υπάρχουν για την διαχείριση των ε, δικαιωμάτων και των συμφερόντων αυτών των τραπεζών και άρα των μετόχων τους. Λοιπόν, ποια είναι τα μέσα για τη διαχείριση της κρίσης από μια, από μια αρχή. Το πρώτο πράγμα είναι η holding η οποία έχει την αρμοδιότητα, τις γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη και την δυνατό. Έχει λοιπόν στοιχεία πολύ ισχυρά και με αυτά μπορεί να διευθύνει τον, τον όμιλο για να διαχειριστεί την κρίση καταλήλως. Είναι δυνατόν λοιπόν μια παρέμβαση αυτού του τύπου να είναι ήδη τώρα σε θέση να επιλύσει το πρόβλημα μέσω τη εξασφάλισης τη εμπιστοσύνη. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Η κρίση που γνωρίσαμε μα ε, έδωσε πολλά να μάθουμε. Εγώ μιλάω για μια διαχείριση κρίση, η οποία ξεκινάει από ένα νόμο από έναν όμιλο και μπορεί να επηρεάσει και άλλους. Δεν μιλάω για μη συστημική κρίση. Εγώ λέω πώς θα αποφύγουμε την κρίση σε έναν όμιλο, σε δύο ομίλους, να μετατραπεί σε συστημική κρίση. Στην πρόσφατη κρίση λοιπόν είδαμε πως οι τράπεζες είχαν ανάγκη από μεσοπρόθεσμη ε, ρευστότητα. Ε, δεν την βρήκα στην αγορά και επειδή οι τράπεζες αυτές είχαν ε, περιουσιακά στοιχεία για να εγγυηθούν την ρευστότητά τους, τη μακροπρόθεσμη, οι οι αρχές δεν είχαν τις ε, αρμόδια μέσα για να πράξουν κάτι τέτοιο. Οι κεντρικές τράπεζε έδωσαν, τέτοια, έριξαν τέτοια αρεστότητα και γι' αυτό και μάλλον δεν έδωσαν την απαραίτητη αρεστότητα και χρειάστηκε να παρέμουν τα κράτη για να χρηματοδοτήσουν ε, μέσω πρόθεσμα τις τράπεζε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα λοιπόν που χρειάζεται να επιλύσουμε. Η πρόταση που κάνουμε είναι η εξή. Να οικοδομήσουμε αυτήν την οντότητα μεσοπρόθεσμα με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου, δηλαδή ένα είδος σύμπραξης. Θα είναι κάτι το οποίο χρησιμεύσει στις, ε, ε, στη σύσταση μιας δομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διαχείριση παρόμοιων φαινομένων. Οι τράπεζα, τράπεζες μάλλον λοιπόν, θα μπορούν στην περίπτωση αυτή να εκδώσουν equity, να ε, τα εγγυηθούν τα κράτη και αυτό, αυτή η αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγει στην, ε, από την αγορά μέσω πρόθεσμη δραστότητα και να αποφύγει την πώληση περιουσιακών στοιχείων για να υπερβεί τις ε, προσωρινές δυσκολίε. Τώρα, αν η κρίση μετατραπεί σε αφαιρεγγιότητα, δηλαδή περάσουμε σε θέση ε, ζημιών, τότε το, αυτή η αρχή θα μπορούσε να συμβάλλει στο να αντιμετωπίσει το κόστος της κρίσης. Εάν τώρα, μάλλον εμείς κάναμε δύο πράγματα. Ε, εάν μάλλον φτιάξουμε την απαραίτητη αρχή και αυξήσουμε τα μέσα, τότε θα έχουμε πετύχει δύο πράγματα. Και θα έχουμε βελτιώσει το moral hazard, ε, την, ε, το να, ε, για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, το moral hazard των τραπεζών υπάρχει μια και μοναδική λύση. Και είναι η μελέτη του τρόπου μια μιας μερικής διάσωσης. Δηλαδή δεν διασώζονται τα πάντα, αλλά διασώζονται τα χρήσιμα. στοιχεία. Λοιπόν, ποια είναι η δυσκολία που υπάρχει για να πετύχουμε αυτήν την ε, προσωρινή μέση κατάσταση, αν θέλετε, μέση διάσωση. Ή, σε μια κανονική κρίση έχουμε το χρόνο να εξετάσουμε την κατάσταση και να κατανοήσουμε την κρίση. Μιλάω για ε, άλλες, ε, οι άλλους τομείς εκτός του τραπεζικού και έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα με τους πιστωτές και να βρούμε μια λύση. Αλλά στην τράπεζα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει διότι η τράπεζα άμα σταματήσει αμέσως καταστρέφει τεράστιες ε, αξίες και εκατομμύρια οικογένειες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα νομικό μέσο με βάση το οποίο θα κατορθώσουμε να συνεχίζεται η τραπεζική δραστηριότητα, να έρθουν σε επαφή οι υπεύθυνοι αυτών των ομίλων, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι οι stakeholders, δηλαδή οι μέτοχοι, έχουν τα δικαιώματα, αλλά υπάρχουν και εμπλεκόμενοι οι οποίοι έχουν υπογράψει άλλου είδους συμβάσεις, άλλου είδους συμβόλαια για συγκεκριμένη περίοδο. Και μπορούν με τον τρόπο αυτό να ικανοποιηθούν οι απαιτήσει τους 30, 40, 50% διότι τότε θα έχουμε δει τι θα μπορεί να διασωθεί. Αλλά αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο. Λοιπόν, το θέμα της ε, υποχρεωτικής ε, εξουσιοδότησης. Ε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι σε περίπτωση κρίσης υπάρχουν εκπρόσωποι αυτών των ενδιαφερομένων, των ε, μετόχων που συνεργάζονται με τις αρχές για να πετύχουν συμφωνίες. Αυτή είναι η μοναδική λύση λοιπόν για να μπορέσει η αγορά να αντέξει περιπτώσεις παρόμοιες χρεοκοπιών. Τελείωσα, μέτρη μου φυσικά στην συζήτηση. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαμάντα. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριο Σον Μάκερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε που με προσκαλέσατε σήμερα. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Οίκων που ακολουθεί και δίνει συνέχεια σε αυτό το σημαντικό θέμα. Τέσσερα σημαντικά θέματα έχω που θα προσπαθήσω με τη σειρά να εξετάσω. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το έργο για τη διασυνορική διαχείριση κρίσεων είναι πολύ σημαντικό και εντάσσεται και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Επίπτωσης. Και έτσι τελικά ένα ενιαίο πλαίσιο συνολικά θα απορρεύσει. Ποιες είναι οι προκλήσεις από τις διασυνοριακές δραστηριότητες πολύ σημαντικό αυτό. Η χρηματοδότηση θα έλεγα ουσιαστικά, όπως και αναφέρθηκε, είναι το κυριότερο στοιχείο. Και τέλει, εν τέλει, πώς θα έπρεπε ένα γενικό ενιαίο συνολικό πλαίσιο να εφαρμοστεί. Στρεφόμενος στο πρώτο ερώτημα αυτό, διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αυτό το οποίο είχα κάνει πριν από την κρίση ήταν <clears throat> ένα τρίλημα χρηματοοικονομικό, ένα τρίγωνο χρηματοοικονομικό με τρεις στόχους χρηματοοικονομική σταθερότητα, χρηματική ολοκλήρωση διασυνοριακά και εθνικές αρχές. Αυτά τα τρία δεν συμπίπτουν. Είναι όπως και το τρίλημα στην χρηματοοικονομική, χρηματονομισματική πολιτική. Λοιπόν, μια επιλογή πρέπει να γίνει. Δύο από τους τρεις αυτούς στόχους μπορούν να συνδυαστούν, όχι όλοι οι τρεις. Και γι' αυτό ένας πρέπει να εγκαταληφθεί. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το status quo, το status quo στην, εσωτερική, στην εσωτερική αγορά, ολοκλήρωση, θέμα εθνικών αρχών, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να είναι σταθερό για το μέλλον θα πρέπει ή να καταλήξουμε σε περισσότερη ολοκλήρωση ή λιγότερη ολοκλήρωση. Στην επόμενη διαφάνεια καθίσταται σαφές αυτό. Η επιλογή ουσιαστικά είναι μεταξύ Α και Β. Επειδή υποθέτω ότι όλοι θα θέλαμε την διασυνοριακή σταθερότητα νομισματικά, χρηματονομισματικά, είναι θα εγκαταλείψουμε τις διασυνοριακές ε, τραπεζικές αυτές ε, μορφές να καταλήξουμε δηλαδή σε εθνικές ε, θηγατρικές... Ε, εταιρείε ε, τι θα γίνει και ότι δεν θα έχουμε μία διασυνοριακή τράπεζα αλλά θα έχουμε μόνο θυγατρικές ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν το τέλος της ενιαίας εσωτερικής αγοράς όμως. Ή η εναλλακτική λύση είναι, και αυτό νομίζω είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, από τις εθνικές αρχές να μεταφερθούμε, να μετατεθούμε στις ευρωπαϊκές αρχές και λύσεις για τα διαφορετικά θέματα του πλαισίου. Εποπτεία, επιτήρηση και ακριβώς ε, αναφέρθηκε αυτό το πρώτο βήμα, ε, ασφάλιση deposits ε, των καταθέσεων και burden sharing, επιμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Να ξεκινήσω φυσικά λέγοντας ότι όλοι ανησυχούμε ιδιαίτερα για το ότι οι φορολογούμενοι έχουν επομιστεί και έχουν πληρώσει τα σπασμένα και πληρώνουν τα σπασμένα και για την πρόληψη κρίσεων σε μεγάλο βαθμό. με τι ανησυχίε των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν πιο πριν και είπαν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πώ μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε την πειθαρχία όσον αφορά τι αγορέ. Δύο θέματα εδώ θα έλεγα. Το πρώτο να μειωθεί η πιθανότητα λαθών και σφαλμάτων. Δηλαδή, να μην μπορεί τόσο γρήγορα να χρεοκοπήσει μια τράπεζα και να υπάρξει και σε σχέση με τα κεφάλαια και τις ε, δράσεις της ε, leverage ratio, μοχλικός, ε, μοχλική αναλογία να γίνει κάτι, καθώς επίσης και υψηλότερα, υψηλότερες απαιτήσει κεφαλαιακές, ώστε να καταλήξουμε σε μειωμένες επιπτώσεις από μια χρεοκοπία να έχουμε δηλαδή τον επομισμό των ζημιών από τον ίδιο τον τραπεζικό τομέα. Το δεύτερο είναι, αν υπάρξει μια τέτοια χρεοκοπία ή αποτυχία, πώς μπορούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Και εδώ έχουμε living wills, το οποίο ως προσέγγιση προσέρχεται στο προσκήνιο. Και από πλευρά των, της λέσχης των 20, G20 αναφέρθηκε. Και σε σχέση με μια πρόταση αντιμετώπισης. Πώς μπορούν δηλαδή οι αρχές να αντιμετωπίσουν τραπεζικές τέτοιες δυσκολίες δυσκολίες τραπεζών. Να αυξηθεί το εύρος των εναλλαγών. Δηλαδή, ή θα χρεοκοπήσει μια τράπεζα ή θα αρχίσει η διαδικασία ε, αυτή και γνωρίζουμε τι συμβαίνει με μια τέτοια μεγαλύτερων διαστάσεων ε, χρεοκοπία ή κλείσιμο μιας τράπεζας. Περνώντας το πιο σημαντικό ε, θέμα, νομίζω το θέμα της ε, διάθεσης κεφαλαίων, funding, εδώ ως οικονομολόγος θα ήθελα να κρούσω κόδωνα κινδύνου. Αν ρίξουμε μια ματιά τριγύρω και δούμε σε σχέση με τις ε, λύσεις που προτείνονται από κάθε ειδικό, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες προτάσεις. Αν τις προσθέσουμε όλες αυτές, έχουμε τεράστιο κόστος για το τραπεζικό σύστημα και θα, οι τραπεζικές υπηρεσίες θα είναι πολύ δαπανηρότερες και ίσως δεν θα υπάρχουν και πιστώσεις που θα είναι δυνατόν να διευκολυνθούν και να διατεθούν. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε τι χρειάζεται και να μην συσσωρεύσουμε σωρευτικά όλες τις προτάσεις τη μία πάνω στην άλλη. Αυτό που θα έλεγα είναι το πιο κατεπήγον είναι, εδώ θα ήθελα να τονίσω το θέμα deposit insurance, ασφάλεια ε, των καταθέσεων. Αν δει κανείς ε, σε σχέση με τις, ε, την ύφεση, κάθε χώρα είχε τις δικές της τέτοιες ασφάλειες για καταθέσεις παραθέσεις. Πράγμα το οποίο ήταν ε, όχι ιδιαίτερα αξιόπιστο και σταθεροποιητικό. Ας δούμε τι έγινε σε σχέση με την Ισλανδία. Δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει επαρκές θα έλεγα πλαίσιο ασφαλιστικό για τις καταθέσεις. Για τις διασυνοριακές τέτοιες συναλλαγές, μια και είναι διασυνοριακές και έχουμε καταθέτες σε διαφορετικά κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχουμε την ασφάλεια καταθέσεων διασυνοριακά, δηλαδή σε ενωσιακό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συμφωνώ με του προλαλήσαντε και του δύο ότι οι τράπεζε θα πρέπει να πληρώσουν τι δαπάνε, Εξάντε δηλαδή εκ προημίου και με βάση πριν όσον αφορά τον πραγματικό κίνδυνο. Μια στρατηγική κινδύνου, αντιμετώπιση κινδύνου. Όταν υπάρχει υψηλό κίνδυνος, υψηλό πριν που καταβάλλεται. Θα έλεγα είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό αν θέλουμε να έχουμε την προσπάθεια ενιαία εσωτερική Χωρί Χωρίς αξιόπιστη ασφάλιση καταθέσεων δεν θα έχουν καταθέσει, δεν θα οδηγούνται σε καταθέσει οι πολίτες μετά από τα όσα έγιναν στην Ισλανδία. Το 2 και το 3 στη συνέχεια. Δύο εναλλακτικέ λύσει για την αντιμετώπιση του ιδίου προβλήματο. Ή upfront ε, θα έχουμε τη δυνατότητα δράση εκ προημίου προληπτικά ή αν πάει κάτι στραβά να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε τα σπασμένα. Να ξεκινήσω με το τελευταίο, το δεύτερο. Τι έχουμε μάθει από την πείρα ότι ποτέ κανένα ταμείο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ε, μεγάλες τράπεζες. Αν δει κανείς ε, τις ΕΠΑ, η FDIC που είναι, έχει καλή ε, κεφαλιακή ε, ροή, για την αντιμετώπιση μεγάλων τραπεζών δεν είναι ικανή. Είναι δυνατόν μόνο σε μικρές τράπεζες να καλύψει ζημιές μέσα σε τρεις μέρες. Μεγάλες τράπεζες δεν μπορούν με τέτοιου είδους ασφαλίσεις ε, να καλύψουν τις ε, ανάγκες και τα σπασμένα. Το ίδιο γίνεται με το Resolution Fund. Μπορούν να αντιμετωπιστούν ανάγκες μικρών τραπεζών. Αλλά σήμερα αντιμετωπίζουμε τα SIFIs, Systemic ε, Important Financial Institutions, συστημικά σημαντικά χρηματοοικονομικά οικονομικά ιδρύματα. Και έτσι λοιπόν αυτό δεν θα ήταν επαρκέ. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και την κυκλική διαμόρφωση τέτοιων ε, ε, γεγονότων. Να δούμε και το θέμα των ε, πριμ, τα οποία θα πρέπει ανάλογα με τον κύκλο αυτό να διαμορφώνονται. Να έλεγα, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με αυτού του είδου τι ασφαλίσει. Να υπάρξει μια αξιόπιστη, αξιόπιστο πλαίσιο ασφάλιση για το burden sharing, επιμερισμό κινδύνων και βαρών, με συγχωρείτε, επιμερισμό βαρών είναι κάτι το οποίο και σε ε, επίπεδο κυβερνήσεων με την Ελλάδα αντιμετωπίζουμε. Το θέμα για το burden sharing και το ανέφερα αυτό δεν είναι ότι κάθε φορά θα πρέπει να είναι έτοιμα κάποια κεφάλαια να βοηθηθείτε, είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί αν χρειάζεται να δούμε πώς θα πρέπει να διατεθούν αυτά τα διαθέσιμα κεφάλαια. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με ένα μικρό βήμα Μικρό βήμα πρώτα. Με αυτά τα living wills πρώτα. Μπορούμε να διοργανώσουμε έτσι, ανα όργανο, ανα το τι θα γίνει με το burden sharing για τις ανάγκες του. Αντί να έχουμε ένα ευρύτατο πλαίσιο burden sharing, να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω εξειδικευμένα να δούμε τι χρειάζεται. Μετά για τις διασυνοριακές τράπεζες και μετά οι μεγαλύτερες τράπεζες, για παράδειγμα για τις τέσσερις ε, σκανδιναβικές χώρες που θα αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις ανάγκες τους. Και τέλος, η το πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων Resolution Fund. Πρώτον, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο Ταμείο Αντιμετώπισης ε, Κινδύνων. Πρέπει να δούμε απλουστευμένα τις ε, δομές. Κάποιες, ε, κάποια τέτοια φαινόμενα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, εμπλέκουν πάνω από χίλιους, χίλια θεσμικά όργανα. Κανείς δεν μπορεί πλέον να κατανοήσει το τι, μπορεί να, τι πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε μια έγκαιρη δυνατότητα παρέμβασης ε, early intervention powers. Λοιπόν, από πλευράς των εμπλεκομένων θα πρέπει το δυνατόν ε, να εμπλακούν το δυνατόν νωρίτερα και να δούμε αν υπάρχει συστημική ή όχι συστημική συνιστόσα που πρέπει να παρέμβουμε, τι μπορεί να διασωθεί και τι πρέπει να χρεοκοπήσει, να αποκοπεί. Και για το συστημικό τμήμα αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων μπορούμε να ε, επιβάλλουμε το συγκεκριμένο εξειδικευμένο σύστημα, ε, πλαίσιο burden sharing, επιμερισμού βαρών με βάση το living will. Και θα ήμουν υπέρ πραγματικά της δεσμευτικής των δεσμευτικών αυτών πλαισίων. Χρειαζόμαστε μια ειδική ε, υπηρεσία, Resolution Agency, για την ε, περίπτωση χρεοκοπιών τραπεζών. Αν υπάρξει τέτοια ε, ενιαία προδιαγραφή σε ευρύτερο πλαίσιο, μπορεί η συνοριακή ε, ε, περίπτωση κρίσεων να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό δεν είναι δυνατόν με memorandum of understandings, με μνημόνια συνεννόησης να λειτουργήσουν όλα αυτά, διότι αυτά δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Αν υπάρχει μια τέτοια κρίση, έκδηλη κρίση, ούτε καν διαβάζει κανείς ένα τέτοιο memorandum of understanding, για να μην πούμε ότι δεν εφαρμόζεται καθόλου βέβαια. Χρειάζεται λοιπόν ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Τελικό ερώτημα. ποιο θα είναι αρμόδιο να παρέμβει σε μια τέτοια κρίση. Ποιο θα δράσει. Και παρότι κανονικά είμαι υπέρ του να έχουμε εξειδικευμένου φορεί και υπηρεσίε για κάτι τέτοιο, θα ήθελα να ακούσω κόδωνα κινδύνου εδώ να μην είμαστε υπέρ της δημιουργίας πολλών, υπερβολικά πολλών νέων υπηρεσιών και φορέων ταυτόχρονα. Κάτι συμφωνώ πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ με τον εισηγητή επ' αυτού. Όμως, εγώ θα έλεγα, ας ξεκινούσαμε με, αυτέ τι αυτές τις νέες supervising authorities, έχουν σημαντικό λόγο να αρθρώσουν και ρόλο να διαδραματίσουν. Σε περίοδους κρίσης η ευρωπαϊκή τέτοια υπηρεσία εποπτείας και επιτήρησης παίρνει τη σκητάλη από την Εθνική Αρχή Εποπτείας Επιτήρησης. Είναι πολύ χρήσιμο. Ας το ενισχύσουμε αυτό. Και ως Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή να δούμε τι πανενοσιακά, πανευρωπαϊκά μπορεί να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο resolution action. δράσης για διάσωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σούμακερ. <clears throat> Ιδιαίτερα όσον αφορά και την τελευταία σας παρατήρηση. Θα λάβει τον λόγο η κυρία Ρίμα, Ρίμα Γιάτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα για να σας μιλήσω για τις απόψεις των τελικών χρηστών. Να πω ότι συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή που ακούσαμε, αλλά θα ήθελα να σας δείξω την άποψη των τελικών χρηστών αποτύχαμε να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και να προστατεύσουμε τους χρήστες του συστήματος. Οι καταθέτες και οι ορισμένοι λιάν επενδύτες έχασαν την εμπιστοσύνη τους γιατί έχασαν καταθέσεις, από αποταμιεύσεις, άλλες επενδύσεις και θεωρούν ότι αυτή η εμπιστοσύνη δεν πρόκειται να επανέλθει εδώ σύντομα. Και η κατάσταση ευχηρετέρευσε όταν διαπίστωσαν ότι οι κυβερνήσεις αποφάσισαν να βοηθήσουν τις τράπεζες. Οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η κατάσταση όπως δημιουργήθηκε ήταν αναπόφευκτη εφόσον δεν υπήρχε κάποιο σύστημα διαχείρισης κρίσεως. Σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαχείριση της κρίσης από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια εφαρμογή για την μείωση του moral hazard και για την μείωση των συστρεβλώσεων της ανταγωνιστικότητας. οι διαδικασίες που υπάρχουν δεν αρκούν για να επιτευχθεί η σταθερότητα. Και επίση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει σε διασυνοριακό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό μια τέτοια επιλογή δεν θα μπορούσε να είναι αποδεκτή ή και επιθυμητή για την εσωτερική αγορά. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα είναι χρήσιμο στην επόμενη κρίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Καταρχάς, με βάση την παγκόσμια φύση του τραπεζικού συστήματος, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν, δυνατό... δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα μηχανισμό έγκαιρης παρέμβασης. Αυτό που θα θέλαμε λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένας τέτοιος υποχρεωτικός μηχανισμός έγκαιρης παρέμβασης θεωρούμε ότι για να είναι αποτελεσματικά κάτι τέτοιο θα πρέπει οι ελεγκτικές αρχές να έχουν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες για να παρεμβαίνουν αρκετά νωρίς στην περίπτωση που έχουμε διασυνοριακή κρίση και η παρέμβαση να βασίζεται σε συμπεφωνημένα εργαλεία τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τι πρέπει να μπορούν να κάνουν οι ηλεκτρικές αρχές. Να αναγνωρίζουν και να προλαμβάνουν την κρίση μέσω του διασυνοριακού ελέγχου των τραπεζικών θέσεων, την εφαρμογή ρυθμιστικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν απαιτήσει για το κεφάλαιο, για τη ρευστότητα, να υπάρχουν ρυθμίσεις που να λειτουργούν ενάντια στον κύκλο και να υπάρχει καλύτερη ποιότητα διαχείρισης. Επίσης δεν θα πρέπει να δρουν μεμονωμένα αλλά σε μακροοικονομικό επίπεδο. Όχι μεμονωμένα και σε μικροεπίπεδο. Από αυτή την πλευρά το σημαντικό είναι η ποιότητα του ελέγχου. Οι ελεγκτικές αρχές και αυτές κάνουν λάθη. Όμως θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ποιότητα, ειδικά στο διασυνοριακό επίπεδο. Δεύτερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο, με το που εντοπίζονται τα πρώτα σημάδια μαλακά ή σκληρά αν θέλετε θα πρέπει να δρούν σε συνεργασία με τις μακροοικονομικές αρχές και να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για σειρά χρεοκοπιών. Θα πρέπει να εντοπίζονται σαφώς ποια θα είναι τα σημεία εκκίνησης αυτών των παρεμβάσεων. Παρακαλούμε Επιβραδύνατε λίγο, ζητάει η Πρόεδρος. Αυτό το σημείο κίνησης μπορεί να ορίζεται μέσω της ε, διάδρασης μεταξύ διαφόρων μικρο και μακροοικονομικών δικτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο και να αφορά θέματα όπως η κεφαλαιοποίηση, η ρευστότητα και το μέγεθος του κινδύνου οι ελεγκτικές αρχές θα επρέχουν τη δυνατότητα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρχές να απαιτούν από ένα ίδρυμα να αυξήσει το κεφάλαιό του, να αλλάξει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, να αλλάζει την διαχείριση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά, διαχείριση της κρίσης. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ex post, εκ των υστέρων, σχεδιασμένοι προκειμένου να ε, μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε εν μέσω της φουρτούνας. Αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούν να περιλαμβάνουν αναστολή της ε, μετατροπής των καταθέσεων σε μετρητά, τους ε, δανειοδότες τελευταίας ευκαιρίας, τις κεντρικές τράπεζες δηλαδή, συστήματα ασφάλισης ε, των ε, καταθέσεων κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, το οποίο δεν θα είναι ούτε υπερβολικά γενναιόδωρο, αλλά ούτε και υπερβολικά στενό. Και θα πρέπει να προχρηματοδοτείτε με βάση ασφάλιστρα που θα βασίζεται στο κίνδυνο και θα είναι γνωστά στους καταθέτες για τις μεγάλες ε, τράπεζες της διεθνής ε, θα πρέπει να υπάρχει ειδική μεταχείριση προκειμένου να έχουμε καλή διαχείριση του συστήματος. Ενδεχομένως ε, να μην αρκεί το σύστημα που ισχύει σήμερα όσον αφορά τις την εγγύηση των καταθέσεων και σίγουρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο καλύτερης και επαρκούς χρηματοδότησης. Τέταρτον, χρήση μέτρων επίληψης κρίσεων. Κάποια ειδικά μέτρα όπως τα living wills, η ζωή διαθήκες αν θέλετε, μπορεί να είναι απαραίτητα για την επίλυση των κρίσεων. Όμως τα living wills θα πρέπει να αναλυθούν πολύ προσεκτικά όσον αφορά τη σχέση κόστους και ωφέλους τους. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η συνέχεια των πληρωμών, η προστασία των καταναλωτών και η ελαχιστοποίηση του κόστους για την κοινωνία. Δηλαδή δεν πρέπει να υπομίζεται το κόστος ο καταθέτης, ο αποταμιευτής, ο φορολογούμενος. Κάτι άλλο. Πρέπει να έχουμε εναρμονισμένους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Ελεγκτικών Αρχών. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα πρέπει να διαθέτει καλό συντονισμό και να έχει αρμοδιότητες απέναντι στις εθνικές αρχές. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της δυνατότητας απόδοσης ευθυνών γιατί αν θέλουμε οι ελεγκτικές αρχές να εγγυώνται την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να υπάρχει και κάποια σαφής εκπροσώπηση των χρηστών στο σύστημα της ελεγκτικής αρχής. Σας ευχαριστούμε πολύ και περνάμε τώρα στην εισηγήτρια, την Ελίζα, η οποία θα ήθελε μάλλον να θέσει κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για όλη τη δουλειά που κάνατε και όλες τις παρεμβάσεις σας. Και σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είναι νομίζω σημαντικό να υποφεληθούμε τα μέγιστα από τη δική σας πείρα και γνώση σε διαφορετικά θέματα. Ένα από τα θέματα είναι ξεκινώντας με το πρώτο πάνελ που θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε αυτό το θέμα είναι ο συσχετισμός μεταξύ εθνικών συμφερόντων και ευρωπαϊκών συμφερόντων. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούμε, να αντιμετωπίσουμε όπως είναι γνωστό. Πώς όμως μπορούμε όταν σταθεροποιούμε, όταν καταλήγουμε σε κοινού κανονισμούς και διατάξεις, πώς μπορούμε στις συμφωνίες που συνάπτουμε σε σχέση με τράπεζες που αποτυγχάνουν στις συναλλαγές τους. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε <clears throat> τα διαφορετικά εθνικά συμφέροντα που εμπλέκονται σε συσχετισμό με διασυνοριακές μεγάλες τράπεζες και συναλλαγές τους. Ποιος είναι ο κανόνας ή η, η προσέγγιση το σώμα των εποπτών, College of Supervisors, είναι αρκετά καλό. Δεν υπάρχει κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, ας το πω να έχει υποδέστερο ρόλο έναντι μεγαλύτερων εμπλεκομένων ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι πτυχές, τι θα γίνει αναόργανο ή θεσμό, ε, institution by institution, τι θα γίνει σε σχέση με τις διατάξεις για τον επιμερισμό των βαρών μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερη ε, στόχευσή μου, να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι το, το, νόημα όλων αυτών των μηχανισμών ως εγχείρημα δεν μπορεί να οδηγεί σε σύγχυση να είμαστε υπέρ των τραπεζών. Όχι. Πρέπει να ελέγχουμε τις ζημιές. Ο έλεγχος των ζημιών και ο η συστημική αντιμετώπιση από πλευρά ελέγχου πιθανών ζημιών. Και όσον αφορά την επιβάρυνση των φορολογουμένων, μείωση του βάρους. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, η δεύτερη παρατήρησή μου, το δεύτερο μου επιχείρημα, το οποίο είναι το ότι εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σύγκληση όσον αφορά την ε, εποπτεία αυτών των θεμάτων που είναι ρευστό ακόμα για ε, ε, ασφαλίσεις καταθέσεων. Όλα αυτά τα ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αποτυχίας ή πριν από αποτυχία έγκαιρα οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά, αυτές τις δυνατότητες για να δράσουν να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, αν υπάρχουν άλλες ε, ε, δυνατότητες πέρα από αυτές τις ασφαλίσεις καταθέσεων για αυτό το στόχο. Ο στόχος της ασφάλισης καταθέσεων είναι να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταθετών. Να μην χρησιμοποιούνται για εκπροημίου κάποιες δράσεις που απαιτούνται και επ' αυτού συμφωνούν όλοι οι προλαλήσαντες. Τρίτο, μπορούμε να πετύχουμε και με ποια βάση μπορούμε να καταλήξουμε και να δημιουργήσουμε αυτά τα εργαλεία, τα μέσα pre-crisis, πριν από την κρίση, να είναι λειτουργικά. Μια και έχουμε τόσο διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, εθνικά, αναχώρα, σε σχέση με τις ε, παρεμβάσεις μας μπορούμε να αναμείνουμε μόνο να εκραγεί ένα πρόβλημα ως έκδηλη κρίση προτού παρέμβει αρμόδια αρχή και προτού δώσουμε μια ειδική ευρωπαϊκή αρμοδιότητα παρέμβασης. Αυτό πρέπει να γίνει, να έχουμε μια έκδηλη κρίση και όπως είπε ο καθηγητής πιο πριν δεν θα πρέπει να σκεφτούμε εδώ την πολυπλοκότητα και τον πολυσχηδή χαρακτήρα ενός τέτοιου καθεστώτος. Πριν γίνει όμως αυτό δεν πρέπει να έχουμε μέσα και εργαλεία που πρέπει να μπορούν να δράσουν σε σχέση με τα δικαιώματα των ε, μεριδιούχων ή εμπλεκομένων σε σχέση με τις διαφορετικές νομικές ε, ε, τάξεις πραγμάτων στις οποίες ζούμε και δρούμε από πλευράς κρατών μελών. Πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν λειτουργικά. Επόμενο θέμα. Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα καθορίζει το τι θα πρέπει να γίνει και πότε ε, triggers, δηλαδή κατόφλια και δράσεις που θα πρέπει με διαφανή χαρακτήρα να μπορούν να λειτουργήσουν αλλά που θα καθορίζουν και τα όρια και την ποιοτική θα έλεγα, τον ποιοτικό χαρακτήρα πληροφοριών που πρέπει να είναι στα χέρια των ρυθμιστών, των ρυθμιστικών αρχών για να μπορούν να δρομολογήσουν δράσεις αποτελεσματικά. Και πιθανότατα τώρα το τελευταίο. Το τελευταίο είναι, μπορούμε να, να έχουμε μια σε τρία επίπεδα ή τέσσερα επίπεδα διαστρωματωμένη δυνατότητα δράσης μεθοδολογικά και συστημικά πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν ε, οι κίνδυνοι έτσι. Ένα άλλο, ε, μια άλλη διάστρωση διασυνοριακών ε, κινδύνων. Ένας άλλος, μια άλλη διαστρωμάτωση εθνικών φορέων ή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τέτοιων συστημικών κινδύνων. Τι μπορεί να γίνει. Και έχουμε εδώ το ε, έμπα ως αρμοδιότητα για την ε, αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων ή τον, το σώμα εποπτών μέσω της έμπα για τις ε, διασυνοριακές δράσεις και τους εθνικούς επόπτες για το εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η δομή που πρέπει να ακολουθηθεί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ομοιογενές πλαίσιο για τις δράσεις όλων, γιατί διαφορετικά δημιουργείται ασάφεια και αβεβαιότητα. Μπορούμε να θεσπίσουμε έναν προσωρινό μηχανισμό ο οποίος θα λειτουργήσει μέχρι ότου καταλήξουμε υστερότερα σε ένα πιο εναρμονισμένο ομοιογενές πλαίσιο. Και τελευταία μου παρατήρηση αν έχουμε ένα μείγμα και με πολλές διασύνδεσεις μεταξύ των διαφορετικών φορέων, αν είχαμε ένα ταμείο αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων, Resolution Fund, θα πρέπει στην διακριτική ευχαίρεια της ΕΜΠΑ ή σε υψηλότερο επίπεδο, μέσα σε ένα κοινό πανενοσιακό πλαίσιο, όπου οι αρμόδιες αρχές για τέτοιες ασφάλειες και θα μπορούν να δράσουν ασφαλιστικό πλαίσιο τραπεζών, να συνέρχονται αυτές και ακόμα αν δοθεί στην ΕΜΠΑ για δράση αυτό το μέσο υπάρχει κάποια κοινή προσέγγιση και συνένεση για την διασύνδεση και αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ όλων αυτών των οργάνων. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Δεν είναι απαντήσεις, είναι περισσότερες, περισσότερα τα ερωτηματικά. Επαρκούμε σε αυτά. Δεν στρέφομαι σε έναν από εσά, αλλά θα ήθελα να καταλήγαμε αν γίνεται σε μια κοινή άποψη μέσω των παρεμβάσεων σας. Ευχαριστώ. Αυτό που, θα... έλεγα να κάνουμε είναι ότι επειδή η συγκήτρια είχε πάρα πολλές ερωτήσεις να μας απαντήσει το πάνελ τώρα σε ερωτήσεις. Παρακαλώ όμως μην εξαντλήσετε όλο το χρόνο που απομένει γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις. Ποιος εξημών θα ξεκινήσει. Θα ακολουθήσουμε την ίδια σειρά όπως και προηγούμενα. Παρακαλώ πολύ σημαντικές ερωτήσεις όλες. Το πρώτο θέμα αφορά το εθνικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον. Πρόκειται, μιλάμε για το ίδιο συμφέρον. Το, το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αυτό όπως και των κρατών, δηλαδή η οικονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Εάν μπορούμε να το πετύχουμε, αν υπάρχει λοιπόν σταθερότητα, τότε οι αγορέ θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Εάν όμω <clears throat> έχουμε κρίση σε οποιοδήποτε επίπεδο εθνικό, ε, τοπικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, φτάνουμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα σας Έχοντα ξεκινήσει λοιπόν μια πολύ σημαντική διαδικασία για τη σύσταση ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, κάτι το οποίο υποστηρίζουμε, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν και οι δυνατότητες και οι ικανότητες των εθνικών εποπτικών αρχών διότι τα εθνικά, τα τοπικά προβλήματα αν δεν επιληθούν σε εθνικό, τοπικό τότε θα μεγεθυνθούν και θα καταστούν ευρωπαϊκά ή και παγκόσμια. Λοιπόν, είναι απαραίτητο λοιπόν ευθύ εξ αρχή να μπορούμε ακόμα και σε τοπικό επίπεδο να επεμβαίνουμε. <clears throat> και τώρα εντάχει. Σχετικά με το συστημικά θεσμικά όργανα πολλές φορές δεν μιλάμε μόνο για συστημικά όργανα αλλά και συστημικές καταστάσεις που μπορούν να προκληθούν όπως η Northern Rock δεν ήταν ένας συστηματικός, συστημικός θεσμός αλλά η κατάσταση η οποία προέκυψε ήταν συστημική Βλέπουμε λοιπόν ότι τέτοιες συστημικές καταστάσει και κινδύνου μπορούν να δημιουργήσουν μη συστημική θεσμή. Υποσχέθηκα πως ε, θα απαντήσω εντάχει. Τώρα κάποια ερωτήματα θα ήθελα να θέσω και εγώ προς τους υπολείπους συναδέλφους μου. Πώς ε, μπορείτε να επιτύχετε την ρευστοποίηση των λεγόμενων θεσμών που είναι λιγότερο συστημική σημασία. Δηλαδή πώς θα έχει η δομή των ευρωπαϊκών χρήματα αγορών εάν αυτή η μη συστημικοί εταίροι, τα μη συστημικά θεσμοί, οι μη συστημικοί θεσμοί θα ε, καταργηθούν. Θα πάψουν να υπάρχουν συστημικά συστημικοί κίνδυνοι. Να απαντήσω λακωνικός θα είμαι. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΕΜΠΑ, η ΕΜΠΑ θα πρέπει να αναπτυχθεί να μεγαλώσει. Τα college αυτή τη στιγμή είναι χώρες που συναντώνται οι αρχές και συζητάνε. Πρέπει να υπάρχουν χώροι για να λαμβάνουν αποφάσεις και η ΕΜΠΑ θα πρέπει να παίξει κυριαρχό ρόλο. Τώρα, δεύτερη ρόλο, τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμεύουν για την αποπληρωμή των χρεών σε περίπτωση αφαιρεγιότητα, όχι. Ε, προτείναμε, εγώ το ταμείο που πρότεινα, γιατί κοιτάξτε, μιλάμε για cross-border group, δηλαδή μιλάμε για ομίλους που έχουν 30, 40, 60 δις ε, ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία. Εντάξει. Αυτοί, οι όμιλοι αυτοί που έχουν χάσει 10 δις χάρη είναι φερέγγοι αλλά δεν ε, λαμβάνουν περαιτέρω χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω πρόθεσμα διότι έχουν περιουσιακά στοιχεία υψηλή ε, αξίας αλλά δεν υπάρχουν ε, οι κατάλληλες δομέ για να αγοράσουν αυτές τα, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να χρηματοδοτήσουν την τράπεζα μέσω πρόθεσμα. Λοιπόν, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Αρχή να αποκτήσει ένα μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορεί να διαχειρίζεται αυτέ τι κρίσει οι οποίε ξεκινούν πάντα ω κρίσει ρευστότητα. Επόμενη ερώτηση. πότε, ποια είναι τα τρίγκε, πότε ξεκινάει αυτή η δραστηριότητα των αρχών. Μα αυτό ε, ε Έγινε στην διακριτική ευχέρεια των αρχών. Θα πρέπει λοιπόν η αρχή να καταλαβαίνει ότι ο τάδε όμιλος ε, αρχίζει να χάνει αξιοπιστία και θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα. Εντάξει, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποιους μηχανισμούς, αλλά εμείς προσπαθούμε να τους ε, γνωρίσουμε αυτούς τους ε, μηχανισμούς έγκαιρα. Τώρα, η ΕΜΠΑ για όλους, νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τους μεγάλους ομίλους. Η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει ένα ισχυρό μέσο. Στην πρόσφατη κρίση, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι πλήρωσαν για την έλλειψη εμπιστοσύνη των αγορών απέναντι στις αρχές. Δεν υπήρχε ευρωπαϊκή αρχή ικανή να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να ε, συστήσουμε έναν τέτοιο, μια τέτοια αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπορέσουμε να ενδεχομένα να προσελκύσουμε και άλλους. Θα σταματήσω πρόεδρε εδώ γιατί βλέπω πως με κοιτάζετε με λίγο βλωσιρώματι. Ο επόμενος. Ευχαριστώ για το θέμα εθνικά συμφέροντα έναντι ευρωπαϊκών συμφερόντων. Μπορούμε να είμαστε απόλυτα σαφείς. Αν δούμε την περίπτωση Φόρτη σε σχέση με τα βελγικά και τα ολλανδικά πράγματα, ήταν θέμα συντονισμού ουσιαστικά. Θα έλεγα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά τις ευρωπαϊκές διασυνοριακές ομάδες πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα default αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Ο πρόεδρος αυτής της αρχής ε, που θα έχει δεσμευτικές εξουσίες είναι πολύ σημαντική υπόθεση για την αποτελεσματική δουλειά, για μια δεσμευτική απόφαση που τότε ξέρουμε όλοι ότι επειδή είναι δεσμευτική όλοι θα συνεργαστούν. Σε περίοδους κρίσης ε, η αρχή αυτή θα έχει αποφάσεις ε, που θα είναι πάνω από τις αρμοδιότητες και εξουσίες των εθνικών αρχών. Πολύ χρήσιμο αυτό. Σε περίοδους κρίσης πρέπει άμεσα, ταχύτατα να λαμβάνονται αποφάσεις. Και ταυτόχρονα στρέφομαι στην τελευταία ερώτησή σας. Αυτό σε σχέση με τις αρχές που θα εμπλέκονται στην κρίση. Αν υπάρχει τράπεζα, μπορεί αφού γίνει η δράση, στη συνέχεια να υπάρξει η επεξήγηση. Πρέπει όμως να υπάρξει πρώτα άμεση δράση. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και EBA, EBA να μπορούν άμεσα να δράσουν, αντί να περιμένουν να δουν, να πληροφορηθούν και να αξιολογήσουν προτού δράσουν άμεσα τι θα γίνει με τις ασφαλίσεις καταθέσεων, deposit insurance. Συμφωνώ θα λέγα με αυτό το οποίο είπατε είπαμε ότι το μη συστημικό τμήμα πρέπει να συρρυκνωθεί, να μειωθεί. Θα πρέπει όμως αυτό να χρησιμοποιηθεί για bailouts, για διάσωση τραπεζών. Θα έλεγα όχι. Εδώ έχουμε το συμφέρον των κατατεθών που πρέπει να διαφυλάστε. Αυτό είναι ο στόχος. Για μεγάλες τράπεζες, όπως είπα πιο πριν, δεν θα υπάρξει αρκετό χρήμα για την κάλυψη τέτοιων αρμοδιοτήτων. Θα διάσει λοιπόν το Ταμείο αυτό ασφάλειας, ασφαλίσεων καταθέσεων για τέτοιε δράσεις όταν θα χρειαστεί να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των καταθετών δεν θα υπάρχουν χρήματα. Άλλο πρέπει να γίνει. Χρειάζεται για τους καταθέτες αυτή, αυτό το κεφάλαιο. Κάτι ξεχωριστό για την αντιμετώπιση και διάσωση τραπεζών. Αυτό πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Μπορεί να γίνει ξεχωριστά. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να συγχαίεται με το άλλο η ασφάλιση των καταθέσεων για τη διάσωση τραπεζών. Μέσα κρίσης εδώ τα νομικά μέτρα είναι παρα... μέσα είναι πολύ σημαντικά. Βλέπω ότι θέλετε να επιταχύνετε, γιατί δεν μπορούμε να ε, χρονοτριβούμε για αυτό το νέο πλαίσιο. Κάποιες χώρες ξεκινούν ήδη με ένα ειδικό πλαίσιο resolution, διάσωσης. Έχει ξεκινήσει ήδη αυτό από κάποιες χώρες. Οι περισσότερες χώρες προβληματίζονται να δουν τι πρέπει να γίνει και έχουν ξεκινήσει οι δράσει. Θα πρέπει να δραχθούμε αυτού του παραθύρου ευκαιρία window of opportunity, να κάνουμε διαφορετικά πράγματα στι διαφορετικέ χώρε, να, να έχουμε παρόμοιες, στόχου που θα α, ακολουθούμε, γιατί διαφορετικά θα έχουμε 27 διαφορετικά καθεστώτα. Χρειαζόμαστε και νομοθεσία για να μπορέσουμε έστω και στο εθνικό επίπεδο προ του ίδιου στόχου να κινηθούμε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τέλο, θα υπάρχουν τρει διαστρωματώσει ή όχι. Πρέπει εδώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο κανόνων, rule book, τι θα γίνεται σε σχέση με συγκεκριμένες ε, ανάγκες και μετά ποιος θα επιληφθεί, ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του έργου. Γιατί πρέπει να είναι σαφή αυτά. Δεν πρέπει σε μια κατάσταση κρίσης να έχουμε ε, συγκεχημένες καταστάσεις. Είναι αναγκαίο να είναι σαφές ε, το πλαίσιο. Τι θα γίνει για τις μικρές τράπεζες, για τις ε, μεγαλύτερες ε, τράπεζες και για τις εθνικές τράπεζες, χώρες τράπεζες. Το ευρωπαϊκό όμως σύστημα το τραπεζικό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Οι κεντρικές τράπεζες κάνουν πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς. Το ίδιο θα συνεχίσουν να κάνουν όμως με βάση τους κανόνες που θα έχουμε από κοινού εκπονήσει. Το σύστημα, συστηματική, ε, το πλαίσιο το οποίο θα διέπει το σύστημα είναι σημαντική υπόθεση. Να έχουμε κοινούς στόχους, κοινούς κανόνες και το θέμα της αποτελεσματικότητας που θα είναι η λιδία λήθος. Και πάνω πάνω στην ακμή του τριγώνου ποιο θα είναι εκείνο, ο οποίο θα παρεμβαίνει αναλαμβάνοντα την αναγκαία δράση όταν θα είναι αναγκαίο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα προκειμένου να σχεδιάσουμε το μέλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα συμφέροντα, αν είναι διεθνή ή ευρωπαϊκά, γνωρίζουμε ότι η σταθερότητα πρέπει να επιτευχθεί σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Πρέπει δηλαδή στο μέλλον να έχουμε κάποια σύγκληση. Δεν πρέπει κάποια μεγάλα μέλη να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα εις βάρος ε, των μικρότερων. Αν θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε σταθερότητα οικονομική και προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να συγκλίνουν τα συμφέροντα όλων. Όσον αφορά τα συστήματα εγγύησης ε, καταθέσεων, συμφωνώ με τον Τιρκ, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες τράπεζες, αλλά όχι αν έχουμε μια μεγάλη χρεοκοπία διασυνοριακών τραπεζών. Δεν νομίζω επίσης ότι αυτό το σύστημα εγγύησης καταθέσεων θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την διάσωση μεγάλων διασυναριακών τραπεζών. Εκεί πρέπει να βρούμε άλλη εναλλακτική λύση. Όσον αφορά τώρα τα triggers, τα σημεία εκκίνησης, είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε έγκαιρες παρεμβάσεις, θα πρέπει να έχουμε κοινού συμπεφωνημένους κανόνες, τόσο ποιοτικού όσο και πισωτικούς. Γιατί ορισμένες φορές οι λόγοι κεφαλαίου προς περιουσιακών στοιχείων είναι δύσκολο να εξεταστούν. Θα μπορούσαμε όμως να βρούμε και άλλα σημάδια έτσι ώστε να έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο ποιοτικών και ποσοτικών σημείων και ενδείξεων. Όσον αφορά τώρα το σύστημα που θα επιλέξουμε, θα πρέπει να επιτρέπει να έχουμε οικονομική σταθερότητα και επίσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ομάδα τραπεζών που εξαιτία της εγγενούς δομής τους πρέπει να ε, ελέγχονται σε τοπικό επίπεδο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ελέγχου και σε εθνικό επίπεδο. Άρα μάλλον ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουμε ένα σύστημα με πολλαπλή διαστρωμάτωση. Όσον αφορά τα ταμεία επίλυσης resolution funds, εγώ θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ελεγκτική Αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητής. Δεν νομίζω ότι μου έχουν κάνει νόημα. Α, τώρα μου κάνουν όλοι νόημα. Λοιπόν, κυρία Χούμπνερ, ευχαριστώ. Ε, δύο ερωτήσεις για τον κύριο Σεν Μάρκερ. Καταρχάς όσον αφορά το ταμείο επίλυσης. Το απορρίπτεται γιατί λέτε ότι κανένα ταμείο δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μία χρεοκοπία μεγάλης τράπεζας. Δηλαδή θα δεχόσασταν αυτό το σύστημα για τις μικρότερες τράπεζες. Και ποιο θα ήταν το κατόφλι σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, ως εμπειρογνώμονας μήπως γνωρίζετε αν έχουν γίνει κάποιες μελέτες αντικτύπου που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και ένα δεύτερο ερώτημα, όσον αφορά τα living wills, τις διαθήκες εν ζωή, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα σχέδιο για τους δύσκολους καιρούς που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τις διασυνοριακές τράπεζες. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτό το διασυνοριακό του θέματος. Οπότε το ερώτημά μου εδώ είναι πώς πιστεύετε ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διασυνοριακή φύση ορισμένων τραπεζών θα αντιμετωπιστούν από τα Living Wills και πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τα ιδρύματα για αυτές τις ε, διαθήκες εν ζωή σε περίπτωση που έχουμε διασυνοριακή δράση. Τέλος, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά αυτά τα living wills, ειδικά όσον αφορά την επενερισμό των ευθυνών, το burden sharing. Επειδή μας μένει μόνο ένα τέταρτο στη διάθεσή μας, θα ακούσω τώρα όλες τις ερωτήσεις. Σφένα, Γιώσεφ Μανουέλα, Τσικλούνα. Όλα. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Νομίζω ότι όλοι μας, η πλειονότητα τουλάχιστον, καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποια ισορροπία μεταξύ της απόλυτης σταθερότητας και της ασφάλειας. Εγώ ως καταναλωτής, επενδυτής και μελλοντικός συνταξιούχος θέλω να έχω κάποιο κέρδος από τις αποταυμιεύσεις μου. Άρα δεν θέλω 100% σταθερότητα γιατί έτσι δεν θα έχω κέρδος. Αυτό που μας λέτε είναι ότι όλες αυτές οι οδηγίες κινούνται προς μια κατεύθυνση ανισορροπίας και θα καταλήξουμε τελικά να μην έχουμε αγορά, να μην υπάρχει ρευστότητα. Μία άλλη ερώτηση. Είναι καλή ιδέα να καταργηθούν κάποια χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Το κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα όχι και τόσο καλά και άλλες χώρες το σκέφτονται. Κατηγορούν για κερδοσκοπία και καταργούν. Νομίζετε ότι είναι καλή ιδέα να καταργήσουμε κάποια προϊόντα. Χρήσιμη ιδέα ή υπάρχουν άλλοι τρόποι έγκαιρης επέμβασης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν. Αυτό το ταμείο που έχει προταθεί για τη χώρα μου, τη Σουηδία, το έχει μελετήσει κανείς, θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό. Εμείς είχαμε αντιμετωπίσει μια κρίση τη δεκαετία του 90 και τα πήγαμε σχετικά καλά, οπότε ίσως αυτό το ταμείο θα ήταν χρήσιμο. Ο κύριος Σον Μάκερ θεωρεί ότι είναι υπερβολικά μικρό και λίγο. Ευχαριστώ για τα σχόλια και ειδικά για το γεγονό ότι ακούμε σχόλια από διάφορες πλευρές. Είναι σημαντικό να έχουμε μία ενιαία κοινή αγορά και βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει προστασία καταναλωτών με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε οποιαδήποτε σύγκληση όσον αφορά το θέμα της εγγύηση των καταθέσεων θα ήταν πολύ καλό. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες. Και αυτό νομίζω ότι βρίσκει πολλούς σύμφωνους και γι' αυτό έχουμε μια καλή βάση από την οποία ξεκινάμε τώρα. Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείται ότι η ύπαρξη μνημονίων ελληλοκατανόησης μεταξύ των κρατών μελών δεν θα επαρκούσαν και θα έπρεπε να έχουμε κάποια άλλη διαδικασία διαχείρισης κρίσεων. Εγώ έχω την εντύπωση ότι τα μνημόνια ελληλοκατανόησης είναι πολύ σημαντικές συμβατικές δεσμεύσεις. Επίσης, αυτή η ελεγκτική η αυτή η αρχή επίλυσης μήπως θα μπορούσε απλά να είναι μια ομάδα από τις ε, ελεκτικές αρχές των κρατών μελών και να μην δημιουργήσουμε δηλαδή μια νέα αρχή εδώ. Και επίσης αυτές οι ελεγκτικές αρχές θα έπρεπε ήδη θεωρώ να συμμετέχουν στην διαδικασία που αφορά την επίλυση των προβλημάτων των, συστημικών ιδρυμάτων. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν κάποια συμμετοχή οι ρυθμιστικές αρχές στο θέμα αυτών των συστημικών ιδρυμάτων. <coughs> Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά τον συσχετισμό ενός σχεδίου εγγύσεων καταθέσεων και λειτουργούντων προγραμμάτων εγγυήσεων εθνικών. Πώς βλέπετε το συσχετισμό τους, ιδιαίτερα σε σχέση με ένα σύστημα που θα αφορά τοπικά ή μόνο εθνικά λειτουργούσες τράπεζες. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα κάποιε πολύ συγκεκριμένες χειροπιαστέ ερωτήσει να διατυπώσω. Αυτή τη στιγμή συζητάμε την αρχιτεκτονική τη χρηματοοικονομικής Ευρωπαϊκή εποπτείας. Εγώ είμαι αρμόδιο για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Όργανο και στην πρόταση έκθεση υπάρχει μια καινοτομία σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου. Η καινοτομία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή θα είχε την εποπτεία εκείνων των οργάνων ευρωπαϊκών επενδύσεων εξορισμού και που θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με διεθνή κριτήρια τα οποία είναι γνωστά. Financial Stability Forum και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο FMI. Αυτή η αρχή θα δρούσε για να μην υπάρχει γραφειοκρατική επιβάρυνση στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω αυτών των εποπτικών αρχών. Αυτοί οι επόπτες όμως θα είχαν τον χαρακτήρα του κατανάθεση επόπτη, κατεντολήν επόπτη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να εξισορροπηθεί αρμοδιότητα και ευθύνη χρηματοοικονομική σε περίπτωση αποτυχίας ή χρεοκοπίας προτείνουμε να υπάρχει ταμείο προχρηματοδοτούμενο σε σχέση με τις, ε, τα έξοδα αυτά που ουσιαστικά ελήφθη υπόψη ακριβώς μέσω της στρατηγικής 2020, 2020 ώστε από πλευράς των χρηματοοικονομικών αυτών φορέων να υπάρξει κάλυψη. Αυτό το ταμείο στην αρχική του μορφή και έχει συζητηθεί αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για δύο πράγματα. Εγγύηση καταθέσεων και διάσωση συστημικά εκείνων των πτυχών που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να διασωθούν. Όταν βλέπουμε σε σχέση με τα σορευόμενα κεφάλαια δεν θα υπαρκούσαν, θα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο να δράσει για την κάλυψη αυτών των αναγκών, όπως το συζητάμε τώρα. Για παράδειγμα, κα, κατ' εξαίρεση ότι αν αυτό χρησιμο, ε, αναγκαίο, θα υπήρχε πρόβλημα, ε, θέμα για την χρήση των κονδυλίων αυτών σε σχέση με τους φορολογουμένους για ένα πλαίσιο Memorandum of Understanding, MOU, για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν αυτά και το πώς θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει σε σχέση με τις διάφορες διαστρωματώσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το Ταμείο έχει το προτέρημα της ε, αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους. Έτσι θα είχαμε και συμμερισμό εκείνων που θα έπρεπε κατά ε, κύριο λόγο να πληρώσουν ε, τις, τα σπασμένα. Και είναι κάτι αυτό που εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να εξεταστεί. Να δούμε τι, θεωρεί, τι θεωρούν οι εισηγητές γι' αυτό, πώς το αντιμετωπίζουν. Θα ζητούσα, Πρόεδρε, επειδή πρέπει να ξεκινήσει μια έκθεση για την Διεθνή ημέρα γυναικών. Αν γίνεται να μου απαντήσουν πρώτα-πρώτα σε αυτή την παρέμβαση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή σε σχέση με το θέμα τραπεζών που θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά μεγάλες ε, σε περίπτωση αποτυχίας για διαρθρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης ε, την, τον διαχωρισμό μεταξύ ε, επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών. Από την άλλη όμως πλευρά, όταν γίνεται λόγος για living wills, εδώ υπάρχει στόχος να διαχωριστούν τα τμήματα εκείνα της τράπεζας που θα επιτρέπονται να αποτύχουν και εκείνων που θα έπρεπε να διασωθούν. Μπορείτε να μας διαφοροποιήσετε, να επεξηγήσετε αυτή τη διαφοροποίηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ επίσης προτιμώ να κάνω λόγο για συστημικούς λόγους και για συστημική προσέγγιση. Γιατί για συστημικούς προσ... Ε, τέτοιους κινδύνους μπορεί οποιοδήποτε, οποιοδήποτε φορέας να, να αντιμετωπίσει. Θα πρέπει συνολικά, σφαιρικά να ε, καλύπτονται αυτές οι πτυχές. Είδα να απουσιάζει μία αναφορά σε σχέση με τις ε, ε, δράσεις αναδιάρθρωσης. Διότι κάνουμε λόγο εδώ για ατομικές ε, δράσεις και προσεγγίσεις, αλλά μπορούν να υπάρξουν και δράσεις αναδιάρθρωσης. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν βρισκόμαστε σε μια κρίση, παράδειγμα. Και είναι προφανώς προφανές ότι υπάρχει μια κλιμάκωση διαφορετικών παρεμβάσεων. Θα έπρεπε να καθοριστεί η πτυχή αυτών. Η μία ομάδα μπορεί να επομιστεί τέτοιες υποχρεώσεις και σε ποιο βαθμό θα ήταν υποχρεωμένη να επομιστεί τέτοιες επιπτώσεις κρίσης. Δεύτερον, μια τέτοια αναδιάρθρωση θα μπορεί να γίνεται σε εθνικό πλαίσιο. Τρίτον, αυτό το οποίο ζητείτε, αν είναι μια αναδιάρθρωση με ένα διαθεσμικό διοργανικό ταμείο ή αν θα έπρεπε με, δημόσιες, ε, ε, ε, με δημόσια κονδύλια να δράσουμε σε κοινοτικό επίπεδο. Κάθε μια από αυτές τις λύσεις ζητεί διαφορετική αντιμετώπιση. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για την αναδιάθρωση Και στο τέλος το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά. Υπάρχει ένα ερώτημα λοιπόν που πρέπει να αποσαφινιστεί εδώ για την, τον εποπισμό του κόστους. Και ποιος θα είναι αυτός. Ο δημόσιος τομέας ο οποίο κάνει αυτές τις πληρωμέ, όταν τις κάνει πρέπει να τις ανακτήσει αυτές τις πληρωμές. Πώς θα γίνει αυτό μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε σχέση με την τρέχουσα κρίση. Πάλι είναι ένα τμήμα το οποίο πρέπει αυτό να το δούμε ξεχωριστά. Την ανάκτηση σε σχέση με το δημόσιο τομέα των πληρωμών που έχουν γίνει για τη σταθεροποίηση του τομέα, του ιδιωτικού αυτού τομέα. Right. Um, I'm sorry you're going to end up with Νομίζω τελικά θα έχετε από 1,5 λεπτό ο καθένα για να απαντήσει ερωτήσει. Ε, συγγνώμη. Να υπενθυμίζω στα μέλη και σε όλου του υπόλοιπου ότι επειδή το απόγευμα έχουμε την ακρόαση με τα εθνικά κοινοβούλια, οι θέσει σα δεν θα είναι ίδιε. Οπότε αν έχετε κάποια έγγραφα να τα πάρετε μαζί σα. Ε, ίσως να αρχίσουμε με αντίστροφη σειρά. Η κυρία Γιάννη θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ να απαντήσω σε εσά δεν υπάρχει καθεστώς ε, το οποίο έχει μηδενικό κίνδυνο αποτυχίας ε, όσες οδηγίες λοιπόν και αν ε, έχουμε για να διασφαλίσουμε 100% την σταθερότητα δεν θα το πετύχουμε. Απλά μειώνουμε τους κινδύνους. Ε, σίγουρα με κάποιο ποσοστό κινδύνου διασφαλίζουμε ανάπτυξη. Αλλά ε, γνωρίζουμε ότι τώρα είχαν ψηλθεί κάποια τοξικά προϊόντα στις χρηματαγορές. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να εξετάσουν πολύ προσεκτικά οι αρχές οι και ίσως η κατάργηση κάποιων προϊόντων ε, μην είναι και ιδιαίτερα κακό. Εγώ ε, γενικά είμαι κατά της ε, κατάργησης κάποιων χρηματοοικονομικών προϊόντων Σε όλη φορά τώρα το Ταμείο Εγγυήσεων των Καταθέσεων, εάν το κόστος αυτό θα το φέρει ο ίδιος ο κλάδος. Τελικά ξέρουμε ότι εν κατακλείδη οι χρήστες είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν και θα περάσει λοιπόν το κόστος στον τελικό χρήστη. Μπορεί να μην συμβαίνει πάντα κάτι τέτοιο, αλλά είδαμε πως μετά την κρίση ότι οι τιμές κάποιων προϊόντων αυξήθηκαν. Μπορεί να υπάρχει μια λύση που θα πρέπει να εξευρεθεί ανάμεσα στις, στον κλάδο και τα κράτη. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει αυτός ο κοινός κίνδυνος ε, να μοιραστεί ανάμεσα στον ε, κλάδο και το κράτος. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση ήταν ε, σχετικά με το Ταμείο εξασφάλισης ε, των καταθέσεων και το ζήτημα μικρών μεγάλων τραπεζών. Όχι, μία της ε, μικρές τράπεζες δεν υπάρχει συστημικό σκήνο και άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει διάσωση. Εάν ε, οι, τράπεζες, οι μικρές τράπεζες χρεοκοπήσουν θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα της post insurance το οποίο θα καταβάλει το κόστος. Θεωρώ πως η διαχείριση της κρίσης είναι ζήτημα που αφορά στις κυβερνήσεις